Pan poseł Tarabella mówi, że powinniśmy zaczynać. Κύριε Ταραμπέλα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Zaczynamy. Άντε κύριε Ταραμπέλα, να ξεκινήσουμε. Συνεχίζεται λοιπόν η συνεδρίαση της Επιτροπής μας να ψηφίσουμε λοιπόν καταρχάς. Γι' αυτό λοιπόν σας είχα ζητήσει και από χθε να φέρετε μαζί τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε πρώτη ψηφοφορία. Μέτρα για την προστασία από α, δυσανιακτώνα. Πρώτη ανάγνωση, έγκριση του σχεδίου. Για δεύτερη ανάγνωση, σύσταση. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό από ό,τι ξέρετε. Και η έγκριση του σχεδίου αυτού θα οδηγήσει σε νέα κανονισμό σε ό,τι αφορά την προστασία των φυτών αυτών. Προετοιμάστηκε λοιπόν από το Συμβούλιο η προτάση αυτή και στη δεύτερη όλα μέλη του Οκτωβρίου θα μπορέσουμε, ελπίζουμε, να την εγκρίνουμε την πρόταση και μάλιστα σε δεύτερη ανάγνωση. Θα ήταν σύσταση για την δεύτερη ενάγνωση. Ηλεκτρονική λοιπόν τώρα η ψηφοφορία. Σας παρακαλώ. Να ψηφίσετε παρακαλώ. Jeśli wszyscy już Εάν ψηφίσατε, δεν ξέρω, έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο και περνάμε στο επόμενο θέμα επενδύσεις, απασχόληση και Ανάπτυξη ε, μεγιστοποίηση των ταμείων επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 16. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η κυρία Νταντσίλα, πρόκειται για μία έκθεση πρωτοβουλίας, κάθε αρμόδια η Επιτροπή περιφερειακή Ανάπτυξης. Και φαντάζομαι ότι η κυρία Νταντσίλα θα μας πει και αυτή δύο λόγια. Για την ε, γνωμοδότηση αυτή, για τις τροπολογίες. Κυρία Νταντσίλα, πάρτε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του κοιότε συζητητέ, όλου του συναδέλφου που κατέθεσαν τροπολογίε, να ευχαριστήσω εδώ και τη γραμματεία για τη δουλειά που έκανε για να έχει έσει τέλος η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι οι επενδύσεις λοιπόν είναι κρίσιμες για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την έκθεση αυτή. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Ε, Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν σας λέμε συγχαρητήρια ακόμα. Να ψηφίσουμε. Τροπολογία υπαριθμών 1. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στο συμβιβασμό υπαριθμών 11. Η ηλεκτρονική παρακαλώ η ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Πέρασε. Εγκρίθηκε παρακαλώ. Ε, εγκρίθηκε ο συμβιβασμό του 11. Συμβιβασμό Α τώρα. Μάλλον συγγνώμη, τροπολογία Α. Πέρασε. Εγκρίθηκε και αυτή η τροπολογία. Η 13 και 14. Υπέρ. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 10. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η υπαρθμόν 9, υπέρ. Υπέρ για την 9. Εγκρίθηκε. Η 10. Η υπέρ, κατά. Απορρίφθηκε. Η 15. Υπέρ. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 20. Υπέρ. Εγκρίθηκε. Η 21. Υπέρ. Εγκρίθηκε. 22. Υπέρ. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για το συμβασμό Β, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 36 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Η 37 Κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 42. Η 42 υπέρ. Όντως. Τη 40, τη 40 πρώτη. Η 42. Υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Για τη 42. Σας ευχαριστώ. πέρασε. Εγκρίνεται. Η 41 υπέρ. Εγκρίθηκε. Η συμβαστική C. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την 41. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ευχαριστούμε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Πολύ ωραία. Συμβιβαστική Συ, λοιπόν, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 43 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Α ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά τι γίνεται με τη 45. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η D, συμβιβαστική D. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 57 υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίθηκε. 58 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 58. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 59 υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίθηκε. Η 60 υπέρ. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Εγκρίνεται. 60 Μάλιστα. Περνάμε στην 64 παρακαλώ. Υπέρ, κατά. Εξταπέντε εγκρίθηκε. Η 66. Αποσύρεται. Μπαίνει το ψυγείο. 67. Υπέρ. Κατά χες, ε, απορρίπτεται. Η 68. Η 68. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 70. Υπέρ. Εγκρίνεται 71 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 71. Κύριε Ντές, είπατε θα υπερψηφίσετε. Αν υπερψηφίσει το ΕΛΚ, εντάξει τι να πω. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 71, έναρξη και πέρας τώρα. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ. 72 υπέρ. Εγκρίθηκε. 73 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Ευχαριστώ. Εγκρίθηκε. 88. Υπέρ. Υπέρ Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 88. Ο κύριος Ντεκάστρο δεν σήκωσε καλά το χέρι του. Να ελέγξουμε την 88 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 88. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 92 υπέρ εγκρίνεται. 93 υπέρ εγκρίθηκε. 97. με την 101. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Άντε, την ελέγξουμε. Κυρία Ανιώ, για την τροπολογία του. Ας την ψηφίσουμε άλλη μια φορά. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Η 99 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ή 100 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική G. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη. Και πέρας τώρα. Εγκρίθηκε. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 109 υπέρ εγκρίθηκε. 110 υπέρ κατά εγκρίνεται. 111 υπέρ εγκρίθηκε. Κυρίε και κύριοι, λοιπόν, τώρα περνάμε στην ε, τελική ψηφοφορία γιατί το κείμενο όπω τροποποιήθηκε. Έναρξη ψηφοφορία, παρακαλώ, για το σύνολο του κειμένου. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε λοιπόν η και τώρα πια μπορούμε να συγχαρούμε την κυρία Νταντσίλα. Συγχαρητήρια. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ψήφο τους και όλα όσα έκαναν για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Όπως ξέρετε το σημείο 13 προβλεπόταν αρχικά για τα υποειδή. Θα συζητούσαμε τα υποειδή, αλλά δεν θα το συζητήσουμε σήμερα. Τώρα έχουμε μία παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΣΑΝΤΕ, από την Κομισιόν, για τους ενδοκρινικούς διαταράχτες ένα θέμα όλος ιδιαίτερος ενδιαφέρον, το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Εξού και το ερώτημα που αποστήλαμε στην Κομισιόν, ή το αίτημα καλύτερα που αποστήλαμε στην Κομισιόν, για να μας διαβιβάσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως ξέρετε. Είναι όμως σημαντικό και για μας, μια και υπάρχει άμεση σχέση με την υγεία την ανθρώπινη. Θα δώσω τον λόγο λοιπόν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος όμως δεν έχει έρθει ακόμα, από ό,τι μου λένε θεωρούσε, υποθέτω, ότι η ψηφοφορία θα διαρκούσε περισσότερο χρόνο. Επομένως, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο θέμα της πανόλης των χείρων. Την Αφρικανική πανόλη των χείρων. Η Γενική Διεύθυνση της ΣΑΝΤΕ θα μας παρουσιάσει για αυτό το θέμα. Ο εκπρόσωπος που θα παρουσιάσει αυτό το θέμα έχει φτάσει άραγε. Δεν έχει φτάσει. Ας περάσουμε τότε στην έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Έχετε λάβει όλες αυτές τις πληροφορίες ε, ηλεκτρονικά, αλλά και σε υπόθεμα χάρτου. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, υιοθετούνται. Επομένως, ή θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε την Κομισιόν ή θα περιμένουμε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτών, θα πιούμε ένα καφέ και μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα θα ξαναρχίσουμε τη συζήτησή μας. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ιδέες, ζητώ συγγνώμη. Προφανώς δικό μου λάθος είναι, γιατί η ψηφοφορία πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Ο κύριος Ταραμπέλα πάντα έχει κάτι να κάνει για να με εκπλήξει. Να με εκπλήξει. Δεν θα σα ξεχάσω ποτέ, κύριε Ταραμπέλα, όταν, ακόμα και όταν φύγω από το κοινοβούλιο. Θα σταματήσουμε λοιπόν, θα κάνουμε μικρό διάλειμμα για 10 λεπτά. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ φταίω δηλαδή, γιατί ουσιαστικά ψήφισαμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν φταίει η Γενική Διεύθυνση Σάντε. Θα κάνουμε λοιπόν 10 λεπτά διάλειμμα.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

θα σας δώσουμε το λόγο λοιπόν χωρίς καθυστέρηση για να ενημερωθούμε για το πρόβλημα αυτό το οποίο μας ε, ενδιαφέρει όλους εταιρεούς. Έχετε το λόγο λοιπόν. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών. Όπως θα ξέρετε σίγουρα, η Κομισιόν παρουσίασε, όπως είχε υποσχεθεί, πριν το καλοκαίρι του 2016, ε, σχέδιο επιστημονικών κριτηρίων για να εντοπίσουμε τους ενδοκρινικούς διαταράχτες στα πλαίσια της εφαρμογής δύο νομοθετημάτων από τη μία την νομοθεσία για την, τα προϊόντα προστασίας των φυτών και την νομοθεσία για τα βιοκτώνα. Στις 15 λοιπόν Ιουνίου η Κομισιόν υιοθέτησε μία ανακοίνωση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που συνοδεύτηκε από μία εκτενή μελέτη αντικτύπου και ενέκρινε ταυτόχρονα δύο σχέδια νομικών πράξεων με κριτήρια για τους κινδύνους με βάση τους οποίους εντοπίζουμε τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Καταρχάς ένα σχέδιο ε, ε, κα, πράξεων για τον κανονισμό και ένα για τον κανονισμό προστασίας των φυτών που θα τα εξετάσουμε στα πλαίσια της διαδικασίας της Πράγας. Όλο αυτό το πακέτο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Κομισιόν, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και να, έχουμε όλα τα κείμενα σε ένα συγκεκριμένο σημείο και όχι διάσπαρτα. Αυτό, είναι, αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε για τα κριτήρια είναι ότι καταρχάς είναι τα ίδια για τα προϊόντα προστασίας των προϊόντων και για τα βιοκτώνα, προστασία συγγνώμη των φυτών. Και για την Κομισιόν το βασικό είναι να έχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας και της υγείας και του περιβάλλοντος. Και σε αυτή την περίπτωση δεν κάνουμε διαφορά. Είτε μιλάμε για βιοκτώνα είτε για προϊόντα προστασίας των φυτών. Επομένως ο, ο σκοπός είναι να εξασφαλίσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας και της ανθρώπινας υγείας και του περιβάλλοντος ε, μέσω και των δύο νομοθετημάτων. Αυτά τα σχέδια κριτηρίων επιστημονικών κριτηρίων πώς δομούνται, σε τι βασίζονται. Καταρχάς, βασίζονται σε τρία στοιχεία με βάση τους τελευταίους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι ε, μια παρενέργεια μετά την έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ε, υπάρχει ένας τρόπος δράσης του διαταράκτη και μια σχέση αιτίου, αιτιατού ανάμεσα ε, στον τρόπο δράσης του ενδοκρινικού διαταράκτη και στην παρενέργεια. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, ορισμένα, με βάση τους ορισμούς του ΠΟΗ. Τα σχέδια κριτηρίων επίσης προσδιορίζουν και τις αρχές οι οποίες θα πρέπει να ε, ακολουθούμε για να εντοπίσουμε τον κίνδυνο. Δηλαδή, θα πρέπει να εξετάζουμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία, ε, ζωικής φύσεως, ε, στοιχεία in vitro και αυτά τα στοιχεία θεωρούμε ότι μπορεί να είναι και σημαντικά για τους ε, ανθρώπους, εκτός και να αποδειχθεί το, αντίθετο. Και θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση με βάση αποδεικτικά στοιχεία. Στη συζήτηση μετά τη δημοσίευση των κριτηρίων, ε, ακούστηκαν ισχυρισμοί ότι τα κριτήρια αφορούσαν μόνο τι γνωστέ επιπτώσει στου ανθρώπου και δεν εφαρμόζαμε παρκώ την αρχή τη προφύλαξη. Όμω, μετά τι ε, εξηγήσει μου και τον τρόπο που τα κριτήρια αυτά σχεδιάζονται, Νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι οι επικρίσεις αυτές είναι αβάσιμες. Επιπλέον, η Κομισιόν προτείνει την τροποποίηση ενός συγκεκριμένου σημείου στο παράτημα των προϊόν, του κανονισμού για τα προϊόντα προστασίας των φυτών για να λάβουμε υπόψη τις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις που έχουμε σήμερα. Αυτή η προτινόμενη αλλαγή βασίζεται στην εντολή που δόθηκε στα πλαίσια του ίδιου καονισμού και η φύση αυτών των τροπολογιών αφορά τις παρεκκλήσεις που υπάρχουν στο πλαίσιο των νομοθετημάτων αυτών και που θα ισχύσουν αυτή τη στιγμή σε εντοπιστεί μια ουσία ως ενδοκρινικός διαταράκτης και θεωρηθεί ενδοκρινικός διαταράκτης. Οι αλλαγές που προτείνουμε λοιπόν είναι να αλλάξουμε την παρέκκληση βασιζόμενη σε αυτό που λέγεται ε, αμεληταία έκθεση σε αυτό το που λέμε ε, αμεληταίο κίνδυνο από την έκθεση. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί, καταρχάς, η εξέταση του κινδύνου θα μας βοηθήσει να εξετάσουμε καλύτερα την, την άλλα υπόψη μας καλύτερα την τρέχουσα επιστημονική γνώση. Επίσης, ε, θα υπάρξει εναρμονισμένη εφαρμογή των κριτηρίων και για τα δύο νομοθετήματα. Γιατί αυτή η έννοια που έχουμε τώρα εισαγάγει για προϊόντα προστασία των φυτών, μια παρέκκληση που θα βασίζεται σε αμεληταίο κίνδυνο από την έκθεση υπάρχει ήδη στα βιοκτώνα, στη νομοθεσία για τα βιοκτώνα. Υπάρχει λοιπόν ευθυγράμμιση πια ανάμεσα στα δύο νομοθετήματα, προϊόντα προστασία των φυτών και βιοκτώνα. Η νομοθεσία ε, για τα βιοκτώνα, το αρχικό της πλαίσιο είναι πιο πρόσφατο από την νομοθεσία προστασίας των φυτών. Και αυτό αντανακλά και την πρόοδο της ε, επιστήμης στη φάση που υιοθετήθηκε το νομοθέτημα για τα διοκτώνα. Η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι τα κριτήρια τα οποία έχει προτείνει είναι πιο επιστημονικά, πιο κατάλληλα από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενδιάμεσα κριτήρια για να εντοπίσουμε τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και μέσω της μελέτης αντικτύπου φάνηκε ότι και τα ενδιάμεσα κριτήρια από καιρού καιρών ε, φτάνουν σε, θετικά, σε ψευδή θετικά αυτό που λέμε ψευδή θετικά. Και δεν μπορούν να εντοπίσουν πραγματικούς ενδοκρινικούς διαταράχτες ακόμα και όταν υπάρχουν. Με τον τρόπο που εφαρμόζονται αυτά τα ενδιάμεσα κριτήρια θεωρούμε ότι είναι κατάλληλα. Και αυτό που προτείνει η Κομισιόν, τουλάχιστον από επιστημονική σκοπιάς, είναι πολύ πιο κατάλληλα για να εντοπίσουν τη σωστή ουσία και να τη χαρακτηρίσουν ενδοκρινικό διαταράκτη. Ε, τα τρέχοντα ενδιάμεσα κριτήρια που ήταν και τμήμα της ε, μελέτης αντικτύπου και της δημόσιας ε, διαβούλευσης που έγινε δεν υποστηρίχθηκαν ούτε από φορείς ενδιαφερόμενους, από stakeholders, ούτε από κάποιο κράτος μέλος. Επομένως, θεωρούμε ότι δεν έχει κανένα νόημα να κρατήσουμε αυτά τα ενδιάμεσα κριτήρια. Η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε τα κριτήρια και να εφαρμόσουμε τα νέα κριτήρια το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν προτείναμε και μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή τους. Τώρα, για να τα πω με μεγαλύτερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά τις επιλογές που είχαμε στην ε, μελέτη αντικτύπου. Μην ξεχνάτε ότι η Κομισιόν δεν προτείνει μια έννοια που θα συμπεριλαμβάνει και κατηγορίες του τι ενδεχομένως μπορεί να είναι ένας ενδοκρινικός διαταράχτης ή υποψή ενδοκρινικού διαταράχτη. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε δεν θα υπάρξουν κανονιστικές συνέπειες για τέτοιες κατηγορίες ενδοκρινικών διαταρακτών. Και θα έχει και νόημα. Δεν θα άξιζε να ορίσουμε τι μπορεί να είναι ενδοκρινικός διαταράκτης. Το βασικό είναι να ορίσουμε τι είναι σίγουρα ενδοκρινικός διαταράκτης και εν τη αυτή περιπτώσει εκεί έχουμε κανονιστικές ε, συνέπειες που απορρέουν από ε, μια τέτοια ταυτοποίηση και ισχύουν. Η Κομισιόν στα επιστημονικά κριτήρια δεν μίλησε για την ισχύ του ενδοκρινικού διαταράχτη, γιατί αποφάσισε να παρουσιάσει κριτήρια για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταραχτών και των κίνδυνων που συνιστούν και η ισχύ τους δεν αποτελεί κριτήριο. Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώθηκε και από πολλούς σημαντικούς επιστήμονες σε μια πρόσφατη συνάντηση που έγινε τον Απρίλιο του 2016. Ήταν μία από τις επιλογές που όμως δεν ακολουθήσαμε κυρίως για επιστημονικούς λόγους. Τώρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τα δύο σχέδια νομικών πράξεων θα υιοθετηθούν με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως σας είπα. Η μία έχει, είναι κατευσιοδότηση πράξη και το άλλο είναι κανονισμός της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά την κατεξιοδότηση πράξης, πράξη, μετά από συζήτηση με τα κράτη-μέλη και τους εμπειρογνώμονές τους κυρίως, θα υιοθετηθεί από την Κομισιόν το κοινοβούλιο, και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ασκήσει έλεγχο. Και το μέτρο για τα προϊόντα προστασίας των φυτών θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην αρμόδια επιτροπή. Και μετά την ψηφοφορία, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα ασκήσει τον έλεγχο. Και τα δύο κείμενα και οι δύο πράξεις θα έχουν κοινοποιηθεί στον ΠΟΗ και εντάσσονται στα πλαίσια του σχετικά νέου κανονισμού του feedback της Κομισιόν. Επίσης, συζητήσαμε και τις δύο πράξεις στα κατάλληλα φόρουμ τον Ιούνιο της Κομισιόν. Τελευταία φορά τα συζητήσαμε την 21η Σεπτεμβρίου και ζητήσαμε τις από τις αντιπροσωπείες να στείλουν γραπτά σχόλια, τα στείλαν και τα αναλύουν αυτή τη στιγμή και την επόμενη συνάντηση με, τα... με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών θα την κάνουμε πριν το τέλος του 2016. επί τη βάση ενός αναθεωρημένου κειμένου που θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα σχόλια που θα έχουν υποβληθεί. Όπως σας έχω ξαναπεί, δίνουμε τεράστια σημασία σε αυτά τα νέα επιστημονικά κριτήρια. Όπως σας είπα, ένας από τους λόγους είναι ότι τα ενδιάμεσα κριτήρια που ισχύουν αυτή τη στιγμή είναι ακατάλληλα. Σκοπεύουμε λοιπόν να προχωρήσουμε με την υιοθέτηση αυτών των νέων κριτηρίων το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη ενός επιστημονικού κειμένου καθοδήγησης για την ε, εφαρμογή των κριτηρίων μαζί με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών και την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων που είναι οι δύο οργανισμοί, οι δύο φορείς που απαιτείται επιστημονικά να εφαρμόσουν αυτά τα κριτήρια για την αξιολόγησή τους, για την αξιολόγηση που θα κάνουν στα βιοκτώνα και στα προϊόντα προστασίας των φυτών. Κλείνοντας, βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε τα κριτήρια αυτά να τεθούν σε ισχύ αμελητή και η απόφαση με βάση τα κατάλληλα επιστημονικά στοιχεία γίνεται ούτω ώστε να έχουμε το καλύτερο επίπεδο προστασία τη ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλοντος. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα κριτήρια που προτείνουμε βασίζονται την καλύτερη δυνατή επιστήμη, στα καλύτερα δυνατά επιστημονικά στοιχεία και τονίζω ότι είναι πρώτη φορά, από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον, παγκόσμια, που κάποια κριτήρια για να εντοπίζουμε τους ενδοκρινικούς διαταράχτες με βάση τα επιστημονικά στοιχεία ενσωματώνται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν η Ευρώπη θα είναι σκαπανέας. Και κατά τη γνώμη μας θα ήταν κρίμα να υπάρξουν οποιασδήποτε καθυστερήσεις σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή. ακούγοντας το διάλογο εδώ στο Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου φαίνεται ότι δεν μας αφορούν σε πολύ τα κριτήρια και το περιεχόμενο γιατί είναι κάτι ασαφές ως πρόταση αλλά ε, πρόκειται περί νομικής ε, διαμάχης μεταξύ, διών, ε, μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου γιατί υπόθηκε ότι η Επιτροπή υπερβαίνει την εντολή της αυτή είναι η μόνη συζήτηση που έχουμε που αφορά το νομικό θέμα και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι πράττει το Συμβούλιο. Αν και αυτοί δίνουν έμφαση στις νομικές συμβουλές, αν έχουν την ίδια άποψη όπως και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, ότι έχετε υπερβεί την εντολή σας και αν θα βγάλετε μια επίσημη ανακοίνωση για να εξηγήσετε και να απολογηθείτε, για να μας εξηγήσετε ότι δεν έχετε πράξει κάτι τέτοιο. Επίσης έχουμε και τις βιομηχανίες και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν αμφιβολίες ε, για αυτή την νομοθετική πρόταση. Αλλά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Αν απορριφθεί η πρότασή σας, τότε θα πρέπει να ε, να διατηρήσουμε τα ενδιάμεσα κριτήρια και ποια θα είναι η επίπτωση αν δεν ε, Υπάρχει ακόμα ένα χειρότερο ε, σενάριο από τα δικά σα τα κριτήρια, αυτό προτείνετε και επίσης να μου πείτε αν δεν είναι σημαντικό να αποσαφηνίσετε καλύτερα το τι αφορά επί τη ουσία αυτή η πρόταση. Κυρία Μούλα, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να βρούμε έναν ορισμό για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες Έχουμε δύο νομικές νομοθετήματα που αφορούν την γεωργία και από πλευρά γεωργίας θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης προϊόντων και να έχουμε και τη δυνατότητα εξαιρέσεων. Έχω αμφιβολίες αν κάνουμε μια αξιολόγηση κινδύνου και ε, να την ε, συμπεριλάβουμε αυτήν στον ορισμό. Θα ήταν πιο σωστό για εμένα να μην ε, δούμε μόνο αυτά τα δύο νομοθετήματα, αλλά και τις διαφορετικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες θίγονται από αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με τα καλλιντικά, με την οδηγία και το νερό. Υπάρχουν διαφορετικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες θίγονται από αυτό το θέμα και θα πρέπει ο ορισμός να ισχύει για όλες το ίδιο. πώς θα χρησιμοποιήσουμε την μελέτη κινδύνου. Και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα στη Γεωργία, γιατί θα πρέπει να καταργήσουμε κάποια διοκτώνα και πώς θα μπορούν να σταματηθούν όλα αυτά ε, στην ε, γεωργία ε, για τη χρήση βιοκτώνων όταν είναι πραγματικά απαραίτητα. Είναι πολύ πρεβλό το θέμα, υπάρχουν πολλοί σχετισμοί, είναι ανοιχτό ερώτημα και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα ώστε να θέσουμε και τα κριτήρια του ΠΟΗ και να τα λάβουμε και αυτά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποσύρει κάποια βιοκτώνα χωρίς ουσιαστικό λόγο. Οτιδήποτε αλλάζει το ορμονικό σύστημα των ανθρώπων θεωρείται ενδοκρινικός διαταράκτης. Ακόμα και τα φαγητά που έχουν βάσει τη σόγια το κάνουν αυτό. Είναι πολλά τα πράγματα όμως που χρειάζομαι. Αν, αν συμπεριλάβουμε και τα φυσικά ιστρογόνα, γιατί αυτά είναι και στην πύρα, στα ε, λαχανάκια Βρυξελών, στην παρακεταμόλη, στον καφέ, είναι τεράστια η λίστα. Το θέμα είναι να πούμε ποιοι είναι οι διαταράκτες, ε, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, όπως καταλαβαίνετε. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες δεν προκαλούν ε, στηρότητα ούτε καρκίνο του μαστού, αλλά είναι δύσκολο να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν ισχύει αυτό. Είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση που α, ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει κάτι ενάντια σε ένα μίασμα. Δεν υπάρχουν όμως αποδεδειγμένα συμπτώματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρα τι, τι ξέρουμε τελικά. το μπενζίλ παράμπεν, το μπενζοπαραμπέν, γνωρίζουμε ότι αυτό ε, έχει, δημιουργεί προβλήματα. Οι γυναίκες παίρνουν συλληπτικά μπορούν τελικά να μείνουν έγιες και τα παιδιά που γεννιούνται δεν ε, δείχνουν κάποια συμπτώματα που έχουν εκτεθεί σε όλα αυτά που περιέχονται στα συλληπτικά και που θεωρούνται ενδοκρινικοί διαταράκτες φυσικά προϊόντα στην ιατρική και που χρησιμοποιούνται στην ε, βιολογική γεωργία είναι εξίσου προβληματικά με τους ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες. Οπότε η αρχή της πρόληψης είναι άχρηστο γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, οποιαδήποτε γενοτομία και θα σταματήσει η παραγωγή ε, προϊόντων, τα οποία όμω τα χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στην ε, βιολογική γεωργία για να μπορέσουμε να παρέχουμε τροφή σε όλο τον κόσμο. Ε, ehm, Είμαι μπερδεμένη γιατί την, τον Ιούνιο που μας πέρασε ασκήθηκε μεγάλη κριτική σε αυτή την πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες η χημική βιομηχανία θα ικανοποιημένη με τα κριτήρια. Ήταν όμως μια μαύρη μέρα για τους ακτιβιστές, αυτούς που συμμετέχουν σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια απόφαση του δικαστηρίου πήρξε ισχυρή κριτική και αν θυμάμαι καλά αν δεν βασίζονται σε μελέτες κινδύνου ε, ρίσκου και άλλε μελέτε επικινδυνότητε, αυτό είναι ένα καλό βήμα. Επίση ε, και ο ΠΟΗ και τα κριτήρια πρέπει, που έχει θέσει πρέπει να διατηρηθούν, να μην υπάρξουν αλλαγέ. Αυτό. Και όταν έχουμε τα αποτελέσματα in vivo και in vitro, ακόμα και σε ζώα, όταν τα έχουμε όλα αυτά, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα βήμα προς την ε, σωστή κατεύθυνση. En daarmee volgens mij de... Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κατεξοδότηση πράξη και αυτό θεωρώ ότι θα αποδυναμώσει τον σκοπό. Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα από πολύ κοντά χωρί να έχω και ένα κείμενο μπροστά μου. Θα θέλαμε να μάθουμε ποιο είναι το οριστικό κείμενο της πρότασης της Κομισιόν και μόνο όταν θα το έχουμε θα μπορούσαμε να πάρουμε θέση πιο ακριβή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Με αφορά το θέμα γιατί είχα καρκίνο και με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αλλά είμαι πολύ προσεκτικός με τις στατιστικές και με τα επιστημονικά πορίσματα που είναι μονόπλευρα. Οι χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής έχουν ε, ε, σε αυτές τις χώρες έχουν αυξηθεί τα ποσοστά καρκίνου γιατί ο καρκίνος συζητείται και με το γύρας. 400 περιπτώσει καρκίνου έχουμε σε 10.000 ε, γυναίκες και 4 ετών, αλλά όσο μεγαλώνει η ηλικία, τα ποσοστά καρκίνου σε μεγαλύτερε ηλικίε είναι πάντα υψηλότερα. Όσον αφορά την φυτοπροστασία, υπάρχει ο κίνδυνος για τους γεωργούς, όμως οι αγρότες στη Γεωργία έχουν κάτω από το μεσόωρο ποσοστό καρκίνου. Όταν είχα εγώ ένα θερμοκήπιο χρησιμοποιούσα πολλά βιοκτώνα όπως και άλλοι γεωργοί και όπως σας είπα είναι κάτω από το μεσόωρο καρκίνο σε αυτή την ε, ομάδα εργαζομένων. Υπάρχουν υποψίες για πολλά προϊόντα θα μπορούσα να απαγορεύσω τα πάντα, τα πλαστικά μπουκάλια, οτιδήποτε. Όμως αυτό που με ενδιαφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει επιστημονική ευθύνη δεν μπορούμε απλώς να απαγορεύσουμε τα προϊόντα φυτοπροστασίας, τα βιοκτώνα χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποια από αυτά πρέπει να απαγορευτούν Ε, γιατί αν ε, δεν το λάβουμε αυτό υπόψη, τότε θα πράξουμε λάθος. Ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική. Είμαι η ίδια αγρότησα και πάνω απ' όλα έχω την υγεία. Νομίζω λοιπόν ότι το πιο σημαντικό για ένα άτομο που ασχολείται με τη γεωργία είναι τα τρόφιμα, τα τρόφιμα τα οποία βάζουμε στο τραπέζι των ανθρώπων τα προϊόντα τα οποία εμείς παράγουμε και οι άλλοι τα αγοράζουν να είναι υγιεινά. Και υπ' αυτή την έννοια η αρχή της προφύλαξης είναι πάνω απ' όλα για μένα. Και είναι σωστό να προσπαθούμε να προστατεύουμε τον κόσμο. Δεν είναι σωστό αντίθετα να δημιουργούμε συνέχεια ε, δυσκολίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Θα πρέπει να θέσουμε τέλος αυτή την αμφιβολία που κυκλοφορεί, σε αυτή την, σε αυτή την εφελώδης ιδέες που κυκλοφορούν γύρω από όλα αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να απαγορευτούν. Ναι, όντω, πρέπει να κάνουμε μια τεράστια συζήτηση και θα πρέπει να βάλουμε στη θέση της τη χημική βιομηχανία, θα πρέπει να συμμορφωθεί με την αρχή της ε, προφύλαξης, θα, πρέπει να σταματήσουν όλοι αυτοί ε, οι βιομηχανίε κτλ. να παράγουν επικίνδυνα προϊόντα. Συχνά, επίσης, οι αξιολογήσεις είναι πειραγμένες. Είναι λάθος, είναι, υπάρχουν, ε, κυκλοφορούν απάτες και δεν είναι σωστό αυτό. Δεν υπάρχουν άλλοι που να θέλουν να πάρουν το λόγο. Μήπως κάποιος θα θέλει να μιλήσει. Όχι. Θα πω λοιπόν ότι ότι εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να ξαναπάρει το λόγο και να απαντήσει στα ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Το ερώτημα που τέθηκε αρχικά για την ομιμότητα της πρότασης θέλω να είμαι σαφής ότι αυτή η ερώτηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου ε, δίνει έμφαση στην ομότητα της απόκλησης, την αλλαγή της φύσης της απόκλησης. Σε αυτό βασίζεται στο risk-based, hazard-based. Άρα δεν, ξέρετε, δεν η νομιμότητα της πρότασης, αλλά του συγκεκριμένου θέματος. Uh, Ήταν πολύ προσεκτική η Επιτροπή για να εξετάσει την νομιμότητα της πρότασης. Πρωτού προχωρήσει, ρωτήσατε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα γιατί δεν έχουμε μπει σε διαβουλεύσεις Είμαστε σε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη ακόμα, με την ε, μόνιμη επιτροπή και το μόνο επιχείρημα που έχουν σε σχέση με την ομότητα συζητήθηκε και η Επιτροπή θεωρεί ότι η φύση αυτού, αυτής της αλλαγής ε, στο παράρτημα είναι απολύτως νόμιμη γιατί μιλάμε για κάποια βασικά στοιχεία. Δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω νομικούς όρους, αλλά η ένδειξη που έχουμε και για την οποία κάνουμε λόγο είναι ότι κάτι που έχει ε, ρυθμιστεί σε ένα παράρτημα ή μέσω, ε, μέσω ενός άρθρου ή μέσω του προημίου τότε αυτό δεν αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο το οποίο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει και η Επιτροπή. Δεύτερον, προφανώς υπάρχει Υπάρχει ενισχύση, ε, ενισχύεται η δύναμη, η ικανότητα της Επιτροπής να προχωράει σε τροπολογίες. Εν ε, επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Αυτό αναφέρεται ότι μπορεί να κάνει τροποποίησεις εν ώψη αυτών των εξελίξεων και θεωρούμε ότι αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση της επιστήμης η οποία εξελίσσεται. Επίσης, ε, η Επιτροπή εξέτασε την ομιμότητα της πρότασης σε σχέση με την τροπολογία για την απόκληση. Η Επιτροπή θα αναλογιστεί και θα σκεφτεί ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος να κάνει αυτή την ε, τοποθέτηση με όσο πιο ολοκληρωμένο τρόπο γίνεται. Άκουσα σχόλια που έγιναν ότι κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση και ότι η πρόταση, ότι η πρόταση στην πρόταση ασκείται πολύ μεγάλη κριτική. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, και να μην καταλήγουμε σε τέτοια συμπεράσματα, γιατί δεν... Ε, ακούσαμε ουσιαστική κριτική που να έχει να κάνει με τα επιστημονικά κριτήρια που έχει θέσει ο Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πω ότι έχουμε 100% συμφωνία, αλλά είναι ευρεία η συμφωνία από ό,τι ακούμε και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και από ε, αγροτικούς κύκλους θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε στην πρόταση υποκατηγορίες Εξήξα τους λόγους που δεν το κάναμε αυτό αλλά παρόλα αυτά αυτή η κριτική η οποία ακούγεται δεν αμφισβητεί την επιλογή των κριτηρίων και τον τρόπο που ε, τα καταρτήσαμε. Υπήρξαν ανησυχίες ότι αυτά τα κριτήρια θα οδηγήσουν σε μια απώλεια ε, πολύ χρήσιμων και ουσιαστικών ε, απαραίτητων προϊόντων. Επιμελώς κοιτάξαμε στην μελέτη δικτύπου αυτό το θέμα και έγινε μια, ένα screening για να έχουμε μια εκτίμηση ε, της κλίμακας των προϊόντων και ουσιών που θα πρέπει που θα, ενδεχομένως θα επηρεαστούν από αυτά τα νέα κριτήρια με βάση τους ορισμούς του ΠΟΗ. Θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική. Το screening δεν είναι η κατάλληλη επιστημονική αξιολόγηση γιατί δεν ήταν όλα τα δεδομένα διαθέσιμα. Επίσης ο χρόνος δεν ήταν αρκετός. Αλλά εκτιμήσουμε ότι 600 περίπου ουσίες και 26 ενδεχομένως να εκπληρούν ε, τα κριτήρια ενός ενεργού συστατικού. Υπάρχει διαφάνεια σε αυτά τα δεδομένα, έχουν ε, ανέβει στην ιστοσελίδα και στη μελέτη αντικτύπου επίσης μελετήσαμε τι θα σημαίνει αυτό και η απόλυτη των προϊόντων για τη γεωργία. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ναι, ε, υπάρχει αντίκτυπος, αλλά προφανώς κάνουμε λόγο για ουσίες με ενδοκρινικούς διαταράκτες, γιατί τα προϊόντα που περιέχουν ε, τέτοιε ουσίε είναι και τα ίδια από μόνο του ενδοκρινικοί διαταράκτε και θα πρέπει να ληφθούν και αυτά ε, υπόψη και να τεθεί προτεραιότητα ως προς αυτά. Έγινε αναφορά επίσης σε φυσικούς ενδοκρινικούς διαταράκτες και αυτό είναι κάτι που επίσης το κοιτάξαμε στη μελέτη αντικτύπου υπάρχουν φυσικοί ενδοκρινικοί διαταράκτες που προκύπτουν, με φυσικό τρόπο από φυτά και που έχουν φυσικές ιδιότητες τα επιστημονικά κριτήρια δεν κάνουν κάτι ως προς αυτό το θέμα, όμως θα επανέλθω στον πυρήνα του ορισμού. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι χρειάζεται να υπάρχουν παρενέργειες. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με ουσίες που δεν δημιουργούν παρενέργειες. Στο παρελθόν, πολλοί από εσάς το γνωρίζετε, υπήρχαν ουσίες οι οποίες είχαν πολύ ισχυρές ε, διατρακτικές ιδιότητες, όπως το DDT, όπου βλέπαμε τις παρενέργειες Ένα, μια συνέπεια ήταν ε, το πώς είχε λεπτύνει το κέλφος από τα αυγά των πουλιών και αυτό μπορούσε να αποδοθεί στις ε, ιδιότητες των ενδοκρινικών διαταρακτών. Αυτός όμως είναι ο πυρήνας της, ε, του ορισμού. Χωρίς παρενέργεια και μια αιτία αιτία του, μια ουσία δεν μπορεί να επιλεγεί ως ενδοκρινικός διαταράκτης. Από την άλλη όμως, και θεωρώ ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν υπάρχουν τέτοιου είδους ουσίες, θα πρέπει και για αυτές να αναλάβουμε δράση, εφόσον έχουμε παρατηρήσει την παρενέργεια. Το δεύτερο βήμα θα ήταν να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή της απόκλησης σε περίπτωση όπου υπάρχει κίνδυνος από έκθεση, από αμέλεια, αν δεν μπορεί να αποδειχτεί κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι η Επιτροπή συμφωνεί. Αυτές οι ουσίες δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην αγορά. Έχουμε εκτιμήσει την κλίμακα και το μέγεθος και τον αριθμό των προϊόντων αυτών που ε, επηρεάζονται από την πρόταση και ισχύει ότι η αρχή της προφύλαξης ε, υπογραμμίζει την ε, πρότασή μας και την νομοθεσία μας και θέλουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον με αυτή την ε, βάση. Όσον αφορά την επίσημη ερώτηση που διέθηκε για την κατεξοδότηση πράξη, αυτό έχει ήδη ρυθμιστεί, έχει καθοριστεί όταν ε, σχεδιάστηκαν οι πρώτες βασικές πράξεις, πότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο για την περαιτέρω εξέλιξη των επιστημονικών ε, κριτηρίων. Το έγγραφο που θέτηκε από την Επιτροπή στις 15 Ιουνίου είναι διαθέσιμο και πιστεύω ότι έχει ανακοινωθεί και στο Κοινοβούλιο είναι κομμάτι του πακέτου που είναι διαθέσιμο μαζί με τη μελέτη δικτύπου και με την ανακοίνωση, άρα μπορείτε να το μελετήσετε. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι η επίπτωση σε άλλες, ε, άλλες κοινωνικές νομοθεσίες, νομοθεσίες. Δεν αφορούν αποκλειστικά ενδοκρινικοί διαταράκτες, ε, τα βιοκτώνα και τη φυτοπροστασία η Επιτροπή στο πλαίσιο της εφαρμογή και σύμφωνα με τις ε, νομικές υποχρεώσεις θα το θέσει και στο πλαίσιο του κανονισμού για τα καλλιντικά. Άρα αυτό αναμένουμε ότι θα γίνει στο μέλλον, θα υπάρξει μια πιο οριζόντια ε, προσέγγιση σε διάφορα αγαθά Καθώς όμως το σύστημα ε, σχεδιάστηκε, ήταν υποχρεωμένη η Κομισιόν να το εντάξει στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα βιοκτώνα και τη φυτοπροστασία. Και αυτό κάναμε σε πρώτη φάση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ε, ε, συμφωνία, ευρύ συμφωνία στους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στα κριτήρια που έχει θέσει, δεν ασκείται κριτική σε αυτά τα κριτήρια και επίσης να τονίσω για αυτός που θέλουν να ψάξουν περισσότερο το θέμα της μελέτης αντικτύπου και υπάρχει διαφάνεια ως προς αυτό ότι να τους πω τα ενδιάμεσα κριτήρια δεν εξυπηρετούν τον σκοπό γιατί έχουμε πολλά ψευδή θετικά τα οποία αποκλείουν κάποια προϊόντα, αλλά για λάθος λόγους. Και παράλληλα δεν επιλέγουν όλους τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που θα επιλέγονταν με τα επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Państwa jest, Υπάρχουν... Ζητείτε λοιπόν το λόγο και υπάρχουν ε, ένα δεύτερος γύρος που προβλέπετε. Ο κύριος Ανιού να πάρει πρώτα το λόγο. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και τους υπόλοιπους ε, που επιθυμούν να πάρουν το λόγο να τον ζητήσουν. Ο κύριο Ανιού, σας ευχαριστώ για τη δεύτερη αυτό γύρο πρόεδρε. Το DDT αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ενδιαφέρον αυτό και κατά δύο τρόπους μάλιστα. Καταρχάς, όταν αφαιρέθηκε, πολλά παιδιά στην Αφρική νόσησαν από αλλονοσία. Άρα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ το, της ζωής των παιδιών και της ζωής της άγρης πανίδας και χλωρίδας. Αν ε, θα απαγορέψουν τον DDT υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα από το οποίο ελοχεύει. Γιατί τα ε, χάπια δυσλεπτικά για τις γυναίκες προκαλούν ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ορμόνες οι οποίες εκλείονται στα ψάρια και άρα θέλουμε να καταργήσουμε τον DDT θα πρέπει να καταργήσουμε και τα αντισυλληπτικά και αναρωτιέμαι τι θα κάνει η κοινωνία χωρίς τα αντισυλληπτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όσο και αν με προκαλεί ο κ. Σακνιό δεν θα σχολιάσω αυτά που είπε. Μία ερώτηση είχα κάνει. για το χρονοδιάγραμμα και την ημερομηνία κατά την οποία θα διατεθεί το κείμενο σε όλους τους ε, φορείς. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε πότε θα μας διατεθεί το κείμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο εκ νέου στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Το κείμενο το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατίθεται και όπως σας είπα βρισκόμαστε στο μέσο της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τη συζήτηση με τους εμπειρογνωμόνες των κρατών μελών για τα βιοκτώνα, για τον, την εφαρμοστική πράξη και ούτω καθεξής. Όπως σας είπα, λάβαμε σχόλια, παρατηρήσεις, ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε και το κείμενο, γιατί θα θέλαμε να μπει μεγαλύτερη σαφήνεια, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Θέλουμε να μην υπάρχουν αμφισημίες, χωρίς φυσικά να τροποποιήσουμε το βασικό στόχο, τη βασική προσέγγιση της πρότασής μας. Και θα ήθελα να τονίζω ότι συμμετέχουν και πρώην εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου στη συζήτηση για τις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Αυτοί λοιπόν έχουν ε, από πρώτο χέρι πληροφορίες για την όλη συζήτηση. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα ρωτήσατε προγραμματίζεται άλλος ένας γύρο συναντήσεων φέτος βάσει του αναφερειμένου κειμένου, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας πω. Δεν νομίζω ότι δηλαδή μπορούμε να ψηφίσουμε το κείμενο αυτό φέτος ακόμα, μέσα στο φετινό έτος. Αυτό φυσικά είναι μια πρόβλεψη δική μου και εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Θα δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα. Νομίζω ότι στις αρχές του επόμενου έτους θα περάσει η εφαρμοστική πράξη. Θέλουμε να περάσουν και τα δύο κείμενα παράλληλα, άρα ελπίζουμε περίπου να το ψηφίσουμε κάπως στις αρχές του επόμενου έτους. Δύο σχόλια τώρα, επιτρέψτε μου, για το DTT, για να διευκρινίσω την ουσία αυτή η οποία χρησιμοποιείται εδώ και μάλλον έχει απαγορευτεί εδώ και πολύ καιρό γιατί ήταν πολλά τα αρνητικά, οι αρνητικές συνέπειες. Η νομοθεσία για το βιοκτώνα και για την προστασία των φυτών. Και οι δύο προβλέπουν μία διάταξη η οποία τι λέει. Αν χρησιμοποιείται, αν χρειάζεται μία ουσία για την καταπολέμηση των διοκτώνων θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση. Τώρα, για το αντισληπτικό χάπι από το στόμα σε ό,τι αφορά τις ε, επιπτώσεις που θα είχε ως ενδοκρινικός τερακτής, συζητήθηκε και στην οδηγία για τα ύδατα και οι εργασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, συνεχίζονται θα ληφθεί υπόψη και λαμβάνεται υπόψη η χρήση του φαρμάκου αυτού στο περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις πληροφορίες αυτές που μας ε, δώσατε και περνάμε στο επόμενο θέμα για την παρουσίαση από τις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά θέματα για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Όπως θα γνωρίζετε, πρόκειται για μία νόσο εξαιρετικά επικίνδυνη, για την οποία προς το παρόν δεν υπάρχει και εμβόλιο. Δεν υπάρχει ε, κίνδυνος για τον άνθρωπο, δεν υπάρχει και μετάδοση σε άλλα ε, ζωικά είδη. Πρόκειται για μία νόσο η οποία πλήττει τους χείρους αποκλειστικά και μόνο. Θεωρείται ε, εξωτική νόσος και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν και κρούσματα στην ε, ε, Ευρώπη, στην Πολωνία ιδιαίτερα. και σε άλλες χώρες. Η νόσος μεταβιβάζεται και περνάει μέσα από τους άγριους χείρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα μας ενημερώσει πιο επακριβώς η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Και ναι, όταν είστε έτοιμοι λοιπόν ε, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ που δίνετε δυνατότητα στην Κομισιόν να εκφράσει την κατάσταση και τις πολιτικές που χρησιμοποιούμε για να περιορίσουμε αυτές τις εξωτικές ασθένειες. Η παρουσίαση θα είναι μακρά, αλλά έχει και οπτικό εδώ υλικό και έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ε, η Αφρικανική Πανόλη των Χειρών υπήρχε και στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε καταφέρει να την περιορίσουμε και να την εξαλείψουμε να την εκριζώσουμε σε ορισμένε περιοχέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι η προσέγγιση μα είναι αρκετά αποτελεσματική σε ό,τι αφορά τον περιορισμό και την εκρίζωση αυτών των εξωτικών ασθενειών. Αυτός που, αυτό που συνέβη πρόσφατα. Ε, θα σας δείξω μια σειρά από χάρτες, οι οποίοι είναι πολύ εύκολοι να τους καταλάβετε, είναι ότι Μιλάμε για ασθένειες των χείρων που δεν επηρεάζουν κανέναν άλλο, κανένα άλλο είδος, ούτε τον άνθρωπο και η οποία μετακινήθηκε από την Αφρική όπου προέκυψε σε μια περιοχή ευρωπαϊκή που είναι ο Κάφκασος. 2007 έγινε αυτό ε, μέσω ε, μεταδοτικού υλικού ας πούμε. Έφτασε στη Γεωργία, βλέπετε τα ποσοστά ε, με μπλε Βλέπετε τον αριθμό των ε, προβληματικών ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μετά άρχισε να φεύγει από αυτή την ε, περιοχή βόρεια, ακόμα πιο βόρεια, το 2011 είχε επεκταθεί σε όλη τη Ρωσική Ομοσπονδία σε διαφορετικές περιοχές Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε το 2011. Μετά η κατάσταση χαλάρωσε λίγο, ηρέμησε λίγο το 2012, αλλά το 2013 προόδευσε η ασθένεια και μπήκε σε μια άλλη χώρα τη περιοχή. τη Λευκορωσία. Και από εκεί Αυτή είναι η εικόνα του 2014. Άρχισε να επηρεάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κατάσταση της προόδου της επιδημίας εδώ τώρα είναι η ρωσική άποψη για το πώς θα είχε συμπεριφερθεί η αρρώστια αν είχαμε εφαρμόσει τις ρωσικές πολιτικές για να περιορίσουμε την αρρώστια. Φυσικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ε, αυτή, είναι από, αυτή η παρουσίαση είναι από μια ρωσική παρουσίαση το 2013. Αυτό που συνέβη στη, στα βόρεια και στην βορειοανατολικά της Ευρώπης είναι ότι το 2014 μπήκε η αρρώστια και όλη τη χρονιά του 2014 κυκλοφορούσε στα σύνορα εκεί, στους, με τους γειτονές μας, Λευκορωσία και Ρωσία. Ε, έχουμε τα, τα κίτρινα ε, που είναι στα, σε άγριους χείρους, ενώ το πράσινο είναι στους α, ήμερους χείρους. Το 2015 επιδεινώθηκε λιγάκι η κατάσταση, αλλά ήταν σχετικά μικρά ο αριθμός των προβληματικών χείρων και ο αριθμό των ε, περιοχών που έχουν επηρεαστεί είναι σχετικά μικρός. Εδώ έχουμε το 2016, είναι ο πιο πρόσφατος χάρτης της αρρώστια και βλέπετε ότι δεν κινήθηκε, δεν μετακινήθηκε η αρρώστια πολύ. Έχουμε περισσότερες τελίτσες ε, γιατί αυξάνουμε την ε, εποπτεία μας και έχουμε και μπλε αστεράκια τα οποία αναφέρονται σε κρούσματα σε ήμερους, εξημερωμένους χείρους. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Συνειδητοποιούμε ότι η περιοχή η οποία έχει πληγεί είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ε, κατάσταση όπως είχε παρουσιαστεί από τα έτη 2007 έως 2014 και είχαμε δει προηγουμένως. Και τώρα ας δούμε την εξέλιξη της αρρώστιας τα τελευταία δύο χρόνια. Μιλάμε τώρα εδώ για το 2015 και εδώ για το 2016. Και βλέπετε η αρρώστια έχει εξαπλωθεί πιο μακριά στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ενώ οι παυλίτσες, τα, τα σύμβολα αυτά, τα κόκκινα και τα πράσινα δείχνουν ε, τους ήμερους και τους, εξημερω, τους εξημερωμένους συγγνώμη, και τους άγριους χείρους ε, και την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άλλος χάρτης εδώ δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων στην περιοχή. Αυτό που είναι ιδιαίτερος ανησυχητικό για μας είναι η κατάσταση στα βόρεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου βλέπετε ένα σύννεφο από πρόσφατες, πρόσφατα κρούσματα που βλέπετε ότι κυκλοφορεί, ε, είναι ενεργός ο ιός, εξαπλώνεται η ασθένεια και στο νότιο πλευρό, στα νότια της Ουκρανίας, δίπλα στη Μολδαβία, έχουμε μια πολύ σοβαρή και ανησυχητική κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μολδαβία πρόσφατα επλήγει από την ασθένεια και μια και είναι μια χώρα γειτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάποιες ανησυχίες για την ικανότητα της χώρας αυτής να περιορίσει την αρρώστια, αποτελεί μια νέα απειλή για μας. Είμαστε συνηθισμένοι βεβαίως στην κατάσταση ε, αυτή, κυρίως στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία, όπου καταφέραμε να περιορίσουμε την κατάσταση, αλλά τώρα έχουμε μια νέα απειλή λόγω της Μολδαβίας. Με δύο λόγια. Ποια είναι η πολιτική μας, ποια είναι τα εργαλεία τα οποία εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία. Να τα διατρέξω γρήγορα. Θα έχουμε το χρόνο να μπούμε πιο βαθιά στη συζήτηση, αν το επιθυμείτε. Καταρχάς, έχουμε πλήρως εναρμονισμένη κτηνιατρική νομοθεσία, ειδικά για τον έλεγχο των ασθενειών των ζώων, των επιζων, Ζωτιών. Έχουμε μία οδηγία του Συμβουλίου, αυτό εκεί αντανακλάνε λοιπόν σε αυτή την οδηγία και έχει κάποιες διατάξεις αυτή η οδηγία για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια. Δύο μείζωνα στοιχεία είναι τα σχέδια κατεπήγοντος όπου τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τα έχουν έτοιμα ούτως ώστε να αναπτύξουν γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσουν την αρρώστια. Το δεύτερο μείζωνα εργαλείο είναι η περιφερειοποίηση θα σας εξηγήσω αργότερα πώς ερμηνεύουμε την αρχή της περιφερειοποίησης. Με δύο λόγια είναι ότι χωρίζουμε την επικράτεια σε δύο τμήματα. Την μολυσμένη, που θεωρείς ότι υπάρχει αρρώστια, και το κομμάτι ας πούμε, της χώρας που δεν έχει κρούσματα. Και το δηλώνεις καθαρό. Η Πολωνία, ας πούμε, βλέπετε ότι είναι χωρισμένη στα δύο. Ένα μικρό τμήμα της Πολωνίας ε, είναι μολυσμένο ε, υπάρχει καραντίνα περιορισμένο και η μεγάλη πλειοψηφία του πολωνικού εδάφους, πολωνικής επικράτειας, είναι και θα είναι καθαρό, χωρίς πανόλη των ε, χείρων. Έχουμε εργαστήρια, τα οποία είναι τα εργαστήρια αναφοράς και παρέχουν υποστήριξη. Και λένε ποια είναι τα διαγνωστικά εργαλεία και τα τεστ που πρέπει να γίνουν, οι δοκιμέ που πρέπει να γίνουν, χρησιμοποιούμε για να συγχρηματοδοτήσουμε και σε ορισμένε περιπτώσει να χρηματοδοτήσουμε 100% κάποια από τα μέτρα για τον έλεγχο των ασθενειών. Έχουμε εποπτεία και προγράμματα εκρίζωση που τα χρηματοδοτούμε με χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κάνουμε εμεί ελέγχου, κάνουμε επιθεωρήσει για να δούμε εάν τα μέτρα όντω χρησιμοποιούνται επί τόπου, ε, όπω έτσι τα έχει σχεδιάσει και φανταστεί ο νομοθέτη, αν όντω γίνονται. Έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, μια ε, ομάδα ε, από κτηνίατρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι έτοιμοι να πάσα στιγμή να αποσταλούν και να πάνε σε οποιαδήποτε χώρα απειλείται ή κινδυνεύει ή παλεύει να περιορίσει την αρρώστια κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δευτερευόντως πάνε και σε ξένες χώρες ε, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι κτηνίατροι, αυτό το team και έχουμε και άλλα εργαλεία που μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αρρώστιες, ε, κατάρτιση, αφύπνιση, μέσω Τη ε, πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για πιο ασφαλή τροφή» ε, έχουμε επιστημονικά στοιχεία, έχουμε τους επιστήμονές μας οι οποίοι μας δίνουν στοιχεία χρήσιμα για την διαχείριση της αρρώστιας. Ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων μας βοήθησε πάρα πολύ για να... και μας έδωσε στοχευμένες επιστημονικές νομοδοτήσει. συνεργαζόμαστε με του γειτονέ μας στα Ανατολικά τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία κυρίω λιγότερο με άλλους γείτονες. Και για, αυτό το, για αυτή τη συνεργασία έχουμε τα πλαίσιο. Βασιζόμαστε σε διεθνεί οργανώσει, όπως ο ΦΑΟ ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζωών και κάτι άλλο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγράμματα ερευνητικά τα οποία έχουν σαν σκοπό να συγκεντρώσουμε νέα μέσα, νέα εργαλεία για να ελέγξουμε τις αρρώστιες. Με αυτά τα πολυάριθμα, όπως βλέπετε, εργαλεία, εφαρμόζουμε αυτές τις γνωστές πολιτικές. Σε περίπτωση που εμφανιστεί μια αρρώστια σε μια γεωργική εκμετάλλευση, έχουμε την νομοθεσία που μας λέει θα κάνετε αυτά. Έχουμε κύκλους, βλέπετε. Ε, 3 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα κτλ. Δυστυχώ για αυτή την αρρώστια πρέπει να σκοτώσουμε, να σφάξουμε τα ασθενή ζώα, το κάνουμε το συντομότερο δυνατό και το ονομάζουμε αυτό εκρίζωση και εφαρμόζουμε περιορισμού σε αυτέ τι ζώνε. Και όταν δεν αρκεί αυτό για να εκριζώσουμε μια ασθένεια μέσα σε ένα-δύο μήνε, α πούμε, τότε πάμε στην περιφερειοποίηση. Όπω σα είπα, αυτή είναι μια αρχή που την έχουμε δεχτεί πια για τον έλεγχο των επιζωτιών. επιζωτιών των, των ζωονόσων. Έχουμε τις ε, περιοχές που είναι μολυσμένες και τις καθαρές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι ο, αυτός είναι ο τρόπος που εφαρμόσουμε την περιφερειοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι, ό,τι είναι γκρι είναι καθαρό. Και οποιαδήποτε επικράτεια είναι χρωματισμένη σε κάποια από τα τρία χρώματα, ε, κόκκινο, ροζ ή μπλε έχει την αρρώστια, παρουσιάζει την αρρώστια και εφαρμόζουμε διαφορετικά μέτρα σε κάθε χρώμα. Η σοβαρότητα των μέτρων έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο, με τον βαθμό του κινδύνου και ο κίνδυνο ε, συνδέεται με την κατάσταση τη αρρώστια. Ε, κόκκινο είναι χάλια. Ροζ είναι ε, καλούτσικο και το μπλε είναι σχετικά ασφαλέ, αλλά όμω υπάρχει αρρώστια παρόλα αυτά. Το κόκκινο είναι όταν ο, η αρρώστια υπάρχει και στου εξημερωμένου και στου άγριου χείρου, ε, ροζ είναι μόνο στους άγριους χείρους και μπλε είναι μια κατάσταση που θεωρούμε προβληματική, αλλά δεν τολμούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η περιφερειοποίηση ε, υφίσταται επικαιροποίηση ανάλογα με την εξέλιξη της αρρώστιας. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση όπου βλέπετε ότι μόνο σε ένα μικρό τμήμα της Πολωνίας, ένα σημαντικό τμήμα της Λιθουανίας και ένα μεγάλο τμήμα της Λετωνίας και ένα τεράστιο τμήμα της Εστονίας, αν όχι όλο, είναι υποπεριορισμό και φυσικά υπάρχει αρρώστια δυστυχώς. Αλλά ε, θέλουμε να το δούμε στη συνολική του προοπτική το θέμα. Παίρνουμε λίγο απόσταση και βλέπουμε ότι η περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιφεροποιείται και θεωρείται μολυσμένη, δεν είναι τόσο μεγάλη σε σχέση με τη συνολική έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κυρίως σε ό,τι αφορά το σύνολο τη ε, χειριάς παραγωγής, τη παραγωγή χειριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι σχετικά μικρό το τμήμα τη Ένωση που ε, είναι μολυσμένο επί τρία χρόνια. Άρα θεωρώ ότι είμαστε μάλλον επιτυχείς ε, στην περιορισμό της νόσου. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την νόσο. Βλέπετε λοιπόν ότι καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να εντοπίσουμε που παρουσιάζονται κρούσματα ακόμα και στα άγρια ζώα. Πάνω από χίλια αγριογούρουν, άγριους χείρους έχουμε θανατώσει τον τελευταίο καιρό και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο αυτό να τα εντοπίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε για τις δραστηριότητες αυτές. Σύγχρονα το δούμε κάποια νομίμα επιλέξιμα μέτρα. Παρατήρηση, παρακολούθηση. Ε, αυτό έχει ως σκοπό να εντοπίζει τα κρούσματα, τη διεξαγωγή ελέγχων, αναλύσεων από ήμερους και άγριους χείρους. Σας τονίζω και πάλι ότι πρόκειται για μία νόσο η οποία απαιτεί μόνο τους χείρους. κάνουμε απολυμάνσεις. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να καταρτήσουμε τους εκτροφείς γιατί αυτή η περιοχή της Ευρώπης ήταν και τόσο μακριά από την Αφρική που ποτέ δεν είχε ζήσει αφρικανική πανόλη των χείρων. Θυμηθείτε την πρώτη μου διαφάνεια. Σε άλλες ε, περιοχές της Ευρώπης ο κόσμος, οι εκτροφείς, οι κτηνίατροι είχαν μια κάποια εμπειρία με την ε, νόσο. Εδώ χρειάζεται μια ευαισθητοποίηση. Γιατί όπως σας είπα, αυτή η νόσος ε, σημαίνει ε, θάνατο για τους χείρους και άρα για να την περιορίσουμε χρειάζεται θανάτωση των μολυσμένων ζώων. Προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό των ζώων που έχουν νοσήσει μέσω σφαγίασης. Εκχωρούμε λοιπόν πόρους, βλέπετε στον πίνακα τη κονδύλια έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τέσσερις ε, χώρες που έχουν σημειώσει κρούσματα τα τελευταία χρόνια. Και εμείς λοιπόν κάνουμε ελέγχους. Έχουμε την διεύθυνση η οποία είναι υπεύθυνη για έλεγχο και για αναλύσεις και τα πορίσματα μας υποδεικνύουν κατά πόσο να πηγαίνουμε καλά ή όχι. Προφανώς τα κρατη τα τέσσερα κράτη-μέλη που έχουν κρούσματα, τα πηγαίνουν αρκετά καλά. αποτρέπουμε αρκετά καλά την ε, εξάπλωση της νόσου. Από ό,τι βλέπετε δεν έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος, όπως είχαν προβλέψει οι Ρώσοι. Δεν έχει πάει στη Γερμανία, για παράδειγμα. Δεν έχει λοιπόν ε, εξαπλωθεί η νόσος γιατί επιβάλλουμε σοβαρούς περιορισμούς ε, στη μετακίνηση που ομολογουμένως είναι οδυνηρή για την βελτίωση της βιοασφάλειας, ε, για τον έλεγχο των μετακινήσεων και φυσικά χρειάζεται και εκχώρηση κονδυλίων. Συνεργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο με το στόχο της ε, περιφερειακής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της νόσου σε διασυνοριακό επίπεδο και δεν μπορούμε να αγνοούμε φυσικά τους γειτονέ μας, πρέπει να συνεργαζόμαστε μαζί τους και γι' αυτό λοιπόν έχουμε ένα γενικότερο οργανισμό στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας. Είναι δική μας η πρωτοβουλία και την προωθούμε, συναντιόμαστε, συζητούμε, συμφωνούμε, προσπαθούμε να εγγυούμαστε την εφαρμογή των μέτρων που έχουμε συμφωνήσει με τους γειτονές μας και γι' αυτό λοιπόν οι εμπειρογνώμονες μας ε, μεταβαίνουν επί τόπου και μας δίνουν από πρώτο χέρι τις εντυπώσεις τους για την κατάσταση. Και αυτό ως τώρα έχει αποτεχθεί αρκετά επιτυχές ως μέθοδος. Σας ομολογώ ότι η συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες έχει βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια. Φυσικά οι προγνώμονες προβαίνουν και σε γνωμοδοτήσεις και συστάσεις και δράσεις που προτείνουν και όλα αυτά φυσικά κοστίζουν χρήματα. αλλά αντιμετωπίζουμε και τα καλά την Υπάρχουν και σημεία κρίσιμα όπου υπάρχουν προβλήματα, γιατί έχουμε και μία νόσο η οποία πλήττει και την εκτροφή αλλά και τα αγριά ζώα. Ένα θέμα είναι το, η χορήγηση τροφής ε, στους χείρους από υπολείμματα της κουζίνας. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται. Ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος που έχουμε εντοπίσει είναι το τι γίνεται με τα κουφάρια των ζώων, των άγριων ζώων που α, πεθαίνουν, που ψοφάνε στα δάση. Και αυτό γιατί τα άγρια ζώα το χειμώνα ε, ενδεχομένως να τραφούν με τα κουφάρια των νεκρών ζώων και αυτό φυσικά ε, μεταβιβάζει, διαβιβάζει την ασθένεια. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε και άλλα προβλήματα στο παγκόσμιο προσκήνιο σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Οι γειτονικέ χώρες μας επιβάλλουν μια οδυνηρή απαγόρευση των εξαγωγών. Η Ρωσία δε, δεν ε, δίνει καν ε, επιστημονική τεκμηρίωση της απαγόρευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει ε, τους χάρτες της περιφερειοποίησης, όπως προβλέπεται και από τα διεθνή πρότυπα και θεωρούμε ότι η απαγόρευση χρήσης των προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το συνόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ήταν δικαιολογημένη. Έγινε και μια σχετική έκθεση από το πάνελ του, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας τον Αύγουστο του 2006 δημοσιεύτηκε. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ακόμα σε φάση αγωγής και φυσικά η Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να αμφισβητήσει την απόφαση της ΠΟΗ. Άρα έχουμε το θέμα και της ασθένειας, έχουμε και θέμα εμπορικό. Ξέρουμε ότι πολλά θα μας βοηθούσαν να καταπολεμήσουμε και να ελέγξουμε την νόσο. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι άγριοι χείροι δεν... Ε, δεν μεταναστεύουν ως είδος. Παραμένουν στην περιοχή τους. Ξέρουμε ότι η βιοασφάλεια είναι η μέθοδος για την αποτροπή μόλυνσης των εκτροφών, των επιχειρήσεων εκτροφής. Αν υπάρχει πρόβλημα κρουσμάτων στην άγρια ζωή, είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση του από την αντιμετώπιση μιας νόσου στις, ε, στους εκροφείς, στις φάρμες, στα αγροκτήματα. Ξέρουμε επίσης ότι η ε, νόσους αυτή δεν έχει φορείς. Δηλαδή, αυτό θα ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο. Αν κάποια δηλαδή, υγιή ε, ζώα ήταν φορείς για μεγάλο διάστημα. Είναι σκληρό ίσω αυτό που θα σα πω, αλλά από την ιατρική άποψη καλύτερα να θανατώνει η ασθένεια η νόσος παρά να συνεχίζει να ζει μέσα σε υγιή ζώα. Και ξέρουμε τι γίνεται λοιπόν και με τους άγριους χείρους. Ξέρουμε ότι υπάρχει Υπάρχουν διάφορε λύσει. Θα μπορούσαμε να είμαστε και πολύ ριζοσπαστικοί. Να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε ε, τα ψόφια ζώα από τα δάση. Και μάλιστα πολύ γρήγορα. Τώρα το πολύ γρήγορα βέβαια είναι σχετικό. Τα ψόφια ζώα αυτά πόσο γρήγορα μπορεί να την εντοπίσει κανεί σε δάσει σε απομακρυσμένε περιοχέ. Υπάρχουν και περιορισμοί πρακτικοί. Αλλά σίγουρα χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση για να αντιμετωπιστεί με βιώσιμο και σωστό τρόπο το θέμα. Άρα, μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ασθένεια και τον πληθυσμό των άγριων χείρων μέσω, για παράδειγμα, στέρηση τροφής και έτσι θα ψοφήσουν τα ζώα αυτά, γιατί ουσιαστικά οι κυνηγοί, οι άνθρωποι είναι αυτοί που παρέχουν τροφή στους άγριου χείρου. ή θα μπορούσαμε να κυνηγάμε και να θανατώνουμε τα θηλυκά, τα οποία αναπαράγονται και έτσι ως εκ τούτου ο πληθυσμό θα μειωθεί σταδιακά για να περιορίσουμε τελικά την ασθένεια. Και τι κάνουμε λοιπόν τώρα τι σκοπεύουμε, μάλλον αυτά ήταν το τι κάνουμε μέχρι τώρα, τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον. Να εφαρμόσουμε τις επιστημονικές αρχές οι οποίες προκύπτουν από την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλισης των Τροφίμων. Το έχουμε συζητήσει και με τους εμπεριογνώμονες και με τους γείτονές μας προς Ανατολάς. Αποφασίσαμε να επιλέξουμε τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση διαχείρισης των χείρων επιλεγμένη ε, και συγκεκριμένη θύρευση των θηλυκών. Αυτό επιλέξαμε. Με πρακτικές που περιγράφονται επακριβώς. Δεν θέλουμε Θέλουμε μάλλον να κάνουμε στοχευμένη θύρευση. Δυστυχώς των ενήλικων θηλυκών. Θέλουμε να απαγορεύσουμε την χορήγηση τροφής στους άγριου χείρου στις περιοχέ αυτέ. Διαφωνούν οι κυνήγοι γιατί δεν θα έχουν φυσικά να κυνηγήσουν το επόμενο, την επόμενη σεζόν. Άρα αντιτίθενται στα κτηνιδευτικά αυτά μέτρα και αυτή η αντιμετώπιση, αυτή η πρόκληση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια σωστή ενημέρωση και συνεργασία προκειμένου να επηρεάσουμε την συμπεριφορά των κυνηγών. Και προσπαθούμε όσο πιο γρήγορα να αφαιρούμε να καθαρίζουμε τα νεκρά ζώα. Με ασφαλή τρόπο. Αυτό φυσικά συνεπάγεται πάλι πόρους και κονδυλία. Και ύστερα έχουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί ήδη έχουμε ένα πρόβλημα με τα ζώα, αλλά τουλάχιστον πρέπει να ενημερώνουμε και τους ανθρώπους. Προσπαθούμε λοιπόν να ενημερώνουμε, να δίνουμε κίνητρα, πόρους, αλλά και κάποια, κάποιους παράγοντες αναστολές. Και προφανώς οι εκτροφείς δεν προτίθονται να κάνουν ότι δεν τους βολεύει και ότι δεν τους αρέσει. Και προφανώς λοιπόν αυτά θα πρέπει να τα ελέγξουμε, θα πρέπει να βελτιώσουμε και την βιοασφάλεια, θα πρέπει οι εκτροφείς να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να ακολουθούν κάποιου κανόνε σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση μια τέτοια νόσου. Και ύστερα έχουμε και την ε, αλληλεπίδραση μεταξύ των εκτροφέων και των κυνηγών. Ιδιαίτερα όταν ένας ε, εκτροφέας είναι και κυνηγό. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Τι κάνω. Φροντίζω τα ζώα μου ή όχι και θα είναι δύσκολος ο χειμώνας για αυτούς. Τι θα κάνουν. Θα προστατεύσουν τα ζώα τους που εκτρέφουν ή θα διασκεδάζουν κυνηγώντα τα Σαββατοκυριακά. Εμείς σκοπεύουμε να επιδείξουμε δυναμισμό. Να προσαρμόσουμε τους κανόνες όπως χρειάζεται και όσες φορές χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά την περιφερειοποίηση, θέλουμε να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται. Βλέπετε και τις περιοχές οι οποίες είχαν πλήχθει και φυσικά σκεφτόμαστε και την ε, στρατηγική εξόδου, το πώς θα σταματήσουν σταδιακά ενδεχομένω αν χρειαστεί αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι είναι οδυνεροί. Αλλά χρειάζεται και κάποια πρόβλεψη για την βιωσιμότητα. στη στρατηγική μας. Είμαστε αρκετά δημιουργικοί και προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τα όρια της ευελιξίας μας. Παράλληλα χρειάζεται και παρακολούθηση, εποπτεία, για να εντοπίζονται τα κρούσματα. Μόνο άμα ξέρουμε που υπάρχουν κρούσματα μπορούμε να προστατεύσουμε τον πληθυσμό των χείρων, την πλειονότητα των χείρων. Πολωνία, Λιθουανία, Λετωνία και δυστυχώς το μεγαλύτερο τμήμα της Εσθονίας έχουν πληχθεί. Έχουν κρούσματα. Αλλά το υπόλοιπο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει παρουσιάσει κρούσματα. Είναι περισσότερο επιστήμη όλα αυτά, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εξαλείφοντας την πυκνότητα των άγριων χείρων δεν εξαλείφουμε την αρρώστια πλήρως, γιατί αυτή η ασθένεια δεν ε, εξαρτάται από τους αγριόχειρους που βρίσκονται στην περιοχή. Ακόμα και αν υπάρχει μια πολύ μικρή ποσότητα αγριόχειρων ε, που έχει ε, ε, πληγεί από την ασθένεια θα παραμείνει η νόσος επειδή παραμένει ζωντανή στα νεκρά, στα, στα νεκρά ζώα και κατά τη διάρκεια του χειμώνου. Βλέπετε εικόνες εδώ είναι μια αργή νόσος. Αυτή ήταν καλύτερα να ήταν γρήγορη, να δρούσε γρήγορα γιατί θα πεθαίνανε μια νυχτή. Είναι όμω μια αργή νόσο όπω είπα. Κάνοντα ε, αυτή τη στενή παρακολούθηση, λέγοντας μας ε, οι άνθρωποι ε, που υπάρχουν ασθενή ζώα, έχουμε 90% εντοπισμό Πρέπει όμως πάντα να φροντίζουμε να αυξάνουμε τη βιοασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα άλλο τρία λεπτά από το χρόνο σας για να σας δείξω μία άλλη νόσο, μία άλλη πιζωτία. Ε, με την άδειά σας θα ήθελα να σας το δείξω και αυτό. Δεν υπάρχουν οι χάρτες βέβαια, απλώς προφορικά θα σας ε, θα σας μιλήσω για αυτή την ε, ασθένεια που την ονομάζουμε στην ε, χώρα μας, στην ε, γλώσσα μας LSD. Είναι μια εξωτική επεισόδια που δημιουργούνται όζοι στο δέρμα των ζώων και αυτή η νόσος πλήττει τα Βαλκάνια και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την Ελλάδα και την Βουλγαρία το Μαυροβούνιο, την Αλβενία, το Κωσυφοπαίδιο και την ε, Φιρόμ. Και ευτυχώ, καταφέραμε να σταματήσουμε δίπλα στην Κροατία και το βόρειο τμήμα της Βουλγαρίας. Άρα η Ρουμανία και η Κροατία είναι ελεύθερη. Πρόκειται για την οζόδη δερματίτιδα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εφάρμοσαν μέτρα τους τελευταίους μήνες με μαζικό εμβολιασμό σε αυτές τις περιοχές. Προσπαθούμε να τη σταματήσουμε. Είναι μια εξωτική ασθένεια η οποία δεν είχε εμφανιστεί προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ άσχημη νόσος, μεταδίδεται με έντομα, δύσκολη περίπτωση και έχουμε τα εργαλεία. Ευτυχώς έχουμε το εμβόλιο το οποίο το χρησιμοποιήσαμε ε, και το χρηματοδοτήσαμε μέσω ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων για εμβολιασμούς και στη Βουλγαρία και στην Κροτία που λειτουργούν σαν προστατευτικό ε, σαν buffer, σαν προστατευτικό προκάλυμα για να μην μεταδοθεί η ασθένεια περαιτέρω και έγιναν και εμβολιασμοί και στις υπόλοιπες ε, περιοχές που αναφέραμε, στην Κοσμοπέδιο, στο Παυροβούνιο, στην Αλβανία, στην Σερβία. Ήθελα να σας πω ότι δεν έχει μεταδοθεί στο βόρα αυτή η νόσος, μόνο στα νοτιοανατολικά είναι γειτονές μας και βασιζόμαστε στην αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης από την πλευρά αυτών των χωρών για να μην μεταδοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Οι ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Ροπέ. Ευχαριστώ που μου δώσετε τον λόγο και ευχαριστώ που συμπεριλάβατε αυτό το θέμα στη σημερινή μερική διάταξη. Στη Λιθουανία και στις χώρες της Βαλτικής η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και δεν βελτιώνεται. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχει βοηθήσει να περιορίσουμε τοπικά το πρόβλημα, αλλά επί της ουσίας έχουμε την εντύπωση ότι, ότι είμαστε σε αναμονή ε, μέχρι να εξαφανιστεί η ασθένεια. Είναι θλιβερή κατάσταση και είναι θλιβερό ε, το γεγονό ότι τα μέτρα που μας βοηθούν αποκλειστικά να περιορίσουμε τοπικά το πρόβλημα, χωρίς όμως να το εξαλείψουμε και οι συμφωνίες που αφορούν ε, στη θρέψη των θηλυκών ε, χείρων δεν έχουν εφαρμοστεί και δεν έχουμε τα κίνητρα για να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, γιατί αυτό θα περιορίσει την αύξηση του πληθυσμού. Δεν είναι σοβαρό μέτρο αυτό, γιατί έχουμε μια σοβαρή απειλή, μια επιζωτία σοβαρή και θα πρέπει να έχουμε δεσμευτικές αποφάσεις, ώστε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Έχουμε νέες συστήσει στην Πολωνία τελευταία και δυστυχώς η κατάσταση ε, γίνεται χειρότερη στην Πολωνία. Μια ελαφριά βελτίωση φαίνεται, διαφαίνεται, όμως είναι μια λάθος εντύπωση αυτή. 20.000 χείρους θανατώσαμε τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή. Και ο λόγος της ύπαρξης του προβλήματος στην ε, συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει εντοπιστεί, δεν ε, καταλάβαμε πώς εισήλθε η νόσο στην περιοχή, ήταν μέσω ζωοτροφής, αν ε, μέσω εντόμων, μυγών, κουνουπιών ή αν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος που μεταδόθηκε η ασθένεια στην περιοχή. Απλώς δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μας θλίβει που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να καταλήξει συμφωνία με τη Λευκορωσία και την Ρωσία. Έχουμε διαφορετικού κανόνε, η δική μα είναι πιο αυστηρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στη Λευκορωσία, παραδείγματο χάρη, μόνο η γεωργική εκμετάλλευση όπου υπάρχει πρόβλημα, μόνο στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν η νόσος να μεταδοθεί από την Λευκορωσία μέσω των ζωοτροφών. Και ένα ακόμα σχόλιο. Πριν από ένα χρόνο περίπου, Έμαθα κάτι σχετικά με τα εμβόλια. Περίμενα να πείτε κάτι για τα εμβόλια. Υπόθηκε και πριν ότι δεν είναι σαφές αν θα παραχθεί το εμβόλιο. Από όσο ξέρω όμως, δεν έχει γίνει ε, προσφορά, δεν έχει γίνει προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία αυτού του εμβολίου. Τι θα κάνουμε λοιπόν στο μέλλον. Πολλοί αγρότες δεν εκτρέφουν χείρους για προσωπικούς λόγους. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γεωργοί αγρότες στην ε, Λουθιουνία που θέτουν αυτό το ερώτημα. Πότε θα μπορέσουν να ανανεώσουμε την ε, εκτροφή χείρων. το κρέας των χείρων χρειάζεται για την εκτροφή. Πότε θα μπορέσουν να είναι σε θέση να ε, συνεχίσουν την εκτροφή. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την αναλυτική έκθεση της λεπτομέρειες που μας έδειξε και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Την εβδομάδα αυτή ήμουνα στη Λετωνία και κατάλαβα πόσο πολύ έχουν πληγεί οι εκμεταλλεύσεις από αυτό το πρόγραμμα και ότι κινδυνεύουν οι αγρότες, κινδυνεύουν να χάσουν τους αβιωτικούς τους πόρους. Θα ήθελα να πω ότι εμείς στη Βαβαρία σκοτώνουμε γύρω στα 60.000 60.000 ε, αγριόχειρους στη Βαβαρία. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτής της νόσου και θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, σοβαροί με τα προγράμματα εξάλληψης. Δεν ξέρω τι γίνεται με την απομάκρυση των ε, πτωμάτων, των ε, κουφαριών των ζωών. Εμείς ξέρουμε ότι με τις ψηλές θερμοκρασίες εξαλείφεται η νόσος. Σίγουρα όμω δεν είναι κάτι απλό. Όσον αφορά για τους λόγους να κάνω κάποιες εικασίε. το να κάνουμε εικασίε για, για τους λόγους δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Αυτό έχει σημασία. Και να κλείσουμε συμφωνίες με τη Ρωσία και θα με ικανοποιήσω πολύ αν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις συμφωνίες γιατί τα προβλήματα στον κλάβο της ε, εκτροφής χείρων είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλο. Όσον αφορά τις τροφές, έχουμε κλειστά συστήματα στα απόβλητα από τα οποία ε, παράγονται ζωοτροφές. Ευχαριστώ ε, για την ενημέρωση που κάνετε για αυτή την οζόδη δερματοπάθεια και σε εμά στην Νότια Γερμανία γνωρίζουμε ότι όλα τα βοηδή πεθαίνουν και αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο εμβόλιο θα ήταν πολύ χρήσιμο να επενδύσουμε κιόλας ώστε να παραχθεί αυτό το εμβόλιο όσο πιο γρήγορα γίνεται Είμαι σε στενή επικοινωνία με τις κλινιτρικές υπηρεσίες και θα ήμασταν πρόθυμοι να βοηθήσουμε στην ε, παραγωγή φαρμάκου, εμβολίου, να διαθέσουμε τα χρήματα για την προστασία των ζώων, της γεωργίας μας, τόσο και για την πανόλη των χείρων, όσο και για αυτή τη νέα ασθένεια, την οζόνη δερματοπάθηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Χάιτουμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και από πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την λεπτομερέστατη αυτή παρουσίαση. Μία ερώτηση από πλευρά ε, των συναδέλφων, του συναδέλφου από τη Φιλανδία. Θα διαβάσω, λοιπόν. Η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων αποτελεί μεγάλη ανησυχία για τους μεγάλου εκτροφείς ε, στην Πολωνία και στι χώρε τη Βαλτική. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αποτρέψουν τη διάδοση και τώρα τα πράγματα είναι υπό έλεγχο και, οι γειτονικές, και στις γειτονικέ χώρες. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αξιόπιστα στοιχεία για την κατάσταση στη Ρωσία και κυρίω στο Σαν Πίτερσπουργκ. Ε, δύο ερωτήσει λοιπόν θα συνάδελφο από την ε, Φιλανδία ρωτάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ μπορούμε να συλλέξουμε πιο, πολύ, πιο πολλά έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία για την κατάσταση στην Λευκορωσία, στη Ρωσία κτλ. Και κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις περιοχές ε, περιορισμού, πώς ε, θα υπάρξει κάποια ανταπόδοση, κάποια αποζημίωση για τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, πλήττονται και τα ζώα τους σφαγιάζονται και μένουν κενές. Και εγώ μία ερώτηση να σας κάνω. Πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση εξάντε μας είπατε για τις ρωσικές αρχές, μας είπατε για την ΠΟΗ και τα σχετικά πορίσματα. Τώρα που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκεχηρίας ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα προσπαθεί να διαπραγματευτεί την κατάσταση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται, για παράδειγμα, το ζήτημα αυτό στο ρωσικό εμπάργο. Ο κύριος Αγνιό. Ευχαριστώ, εξαιρετική παρουσίαση, πολύ ενημερωτική, πολύ σας ευχαριστώ. Για τα συμπτώματα να ρωτήσω. Τα συμπτώματα είναι... Ε, περνάνε παρατηρήτητα για κάποιο χρονικό διάστημα και ε, από την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι την, ε, το θάνατο του ζώου, πόσο καιρός περνάει γιατί αυτό έχει σημασία. Και φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους αγρίους χείρους ε, είναι καθοριστική σε ό,τι αφορά τη μετάδοση της ασθένειας. Δεν έχουμε πολλές δυνομένο Βασίλειο. Έχουν εκλείψει τα τελευταία 50 χρόνια. Ωστόσο υπάρχει εκτροφή και κάποια ζώα έχουν τραπετεύσει και έτσι πλέον έχουμε πάλι κάποιους αγριόχειρους. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλά ε, ζώα, πολλά γουρουνιά τα οποία τα εκτρέφουν σε εξωτερικούς χώρους όπου θα είχαν ενδεχομένως επαφή με τους αγριόχειρους. Και αυτό ενδεχομένως ε, θα ήταν προβληματικό. Άρα προσπαθούμε να δούμε πώς ε, θα μπορούσε να γίνει η διάδοση πέρα από τη μετακίνηση των χείρων και την κατανάλωση των κουφαριών, το οποίο ελέγχεται σχετικά εύκολο. Επίσης, ε, τι γίνεται με τα πουλιά, τα αρπακτικά πουλιά, τους γήπες ε, που ενδεχομένως στρέφονται από τα κοφάρια και μετά μεταναστεύουν. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα μετάδοσης, γιατί είδαμε ότι η γρήπη των πουλερικών, για παράδειγμα, μεταδόθηκε από τα μεταναστευτικά πουλιά. Όταν μιλάτε για τη Ρωσία, δεν λέω ότι διαφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά μου φαίνεται ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται και μάλλον υπεύθυνα απαγορεύοντας τις εξαγωγές. Εμένα μάλλον υπεύθυνη αντιμετώπιση μου φαίνεται αυτή. Παρ' όλα αυτά, οι παγκόσμιες αρχές βγήκαν και είπαν ότι λάθος ήταν η κίνηση. Ίσως και να μην καταλαβαίνω καλά, για πείτε μου όμως. Και τέλος, κάνατε μια πολύ εύστοχη παρατήρηση για όσου που εκτρέφουν παράλληλα χείρου και κυνηγούν αγριό παράλληλα. Και έχουμε και κάποιους, ε, για να τα μεταφέρω στα πολυρικά, ε, στην πατρίδα μου το θέμα αυτό, που έχουν ε, και εκτρέφουν πουλερικά και κυνηγούν φασιάνου παράλληλα. Και έχω και ένα συγκεκριμένο υπόψη μου εδώ πέρα. Ευχαριστώ κύριε obrigado. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες για τη Σαρδινία, παρακαλώ, που ανήκει στην Ιταλία και όπου υπάρχει η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Στην Ιταλία είναι ενδυμική η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Ε, διερωτώ με, ή έγινε κάποια επιμόλυνση. Έχετε καμία ιδέα γιατί ξέσπασαν αυτά τα κρούσματα στην Σαρδινία που είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Επίσης, σε ορισμένε χώρες Υπάρχει πολύ αυστηρή νομοθεσία που ζητάει εξωτερική, απαιτεί εξωτερική αξιολόγηση και μπορεί να θεωρήσουμε ότι μία περιοχή τουλάχιστον 100 τετραγωνικά μέτρων ως ημικαθαρή, γύρω από μία γεωργική εκμετάλλευση δηλαδή. Υπάρχει δηλαδή μια ζώνη μαξιλάρι ανάμεσα στα, στους εξημερωμένους χείρους και τους αγριόχειρους. Με αυτόν τον τρόπο δεν έρχονται σε επαφή ε, οι αγριόχειροι με εξημερωμένους χείρους. Ε, χάρη σε αυτές, σε αυτές τις περιοχές μαξιλαράκια ας πούμε. Διερωτόμαστε γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος σε περισσότερες χώρες. Για αυτές τις εστίες, ε, σε αυτές τις χώρες Υπάρχει η σκέψη να γίνουν κάποιες επενδύσεις σε μια τέτοιου είδους υγειονομική προφύλαξη, ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί το βασικό πρόβλημα που είναι η επαφή ανάμεσα στους αγριόχειρους και στους εξημερωμένους χείρους. Δηλαδή, Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, περιοχές κινδύνου, ποιες είναι ακριβώς οι περιορισμοί για τα ζώα τα οποία μεταφέρονται από τις, γεωργικές, ε, από τις ε, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα σφαγεία. Τι κάνετε, ελέγχετε όλα τα ζώα ή δειγματοληπτικά τα ελέγχετε. Και επίσης, για ζώα τα οποία προέρχονται από μολυσμένες περιοχές. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αγριόχειρους. Μπορούμε να έχουμε και ξημερωμένους χείρους που είναι άρρωστοι. Γιατί Ξέρουμε πολύ καλά, ας πούμε, ότι ο, ο ιός υπάρχει και στο, και στο κρέας, αλλά και στα μεταποιημένα προϊόντα από άρρωστα ζώα. Θέλω να ξέρω, λοιπόν, ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι περιορισμοί που προβλέπετε για να μην διαδοθούν και να μην να τεθούν σε κυκλοφορία τέτοια προϊόντα. Επίσης, Ποια είναι τα μέτρα υγειονομικής επαγρύπνησης που έχετε ενεργοποιήσει ούτω ώστε να εξασφαλίσετε ότι αυτή τη στιγμή σκοτώνουμε τα ζώα και τα ξανα... και, και ξαναγεμίζουμε ας πούμε αυτές τις ε, εγκαταστάσεις δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στις, α, στους αγριόχειρους και στους εξημερωμένους χείρους. Επίσης κάτι άλλο, η κλασική πανόλη των χείρων, όχι η αφρικανική. Ε, η κλασική πανόλη των χείρων ε, έχει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με την αφρικανική πανόλη των χείρων, μόνο που η εξέλιξή της είναι πολύ πιο γρήγορη. Επομένως θα πρέπει να γίνεται μια σαφής διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις δύο αρρώστιες ε, που έχουν τα ίδια συμπτώματα αλλά είναι διαφορετικές. Ε, είναι και οι δύο σοβαρές, έτσι. Και οι δύο υπόκεινται σε σχέδια εκρίζωσες, όμως για την κλασική πανόλη των χείρων υπάρχει το εμβόλιο. Παρότι ας πούμε, το να καταφύγουμε στο εμβόλιο ε, είναι σαν να ομολογούμε ότι δεν μπορούμε να εκριζώσουμε την αρρώστια. Αλλά τι να κάνουμε, τουλάχιστον να κάνουμε αυτό. Και το τελευταίο μου ερώτημα αφορά το εμπάργκο, δηλαδή την δυνατότητα να επιτρέψουμε χώρε οι οποίες δεν έχουν πληγεί από την αφρικανική πανόλη των χείρων να μην πληγούν από εμπάργκο για τα προϊόντα τους. Να μην θεωρηθεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα πράγμα. Μην τα βάλουμε όλα τα προϊόντα της Ευρωπαϊκή Ένωση στο Γιοκαζάνι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση που μας έκανε. Υπήρχαν πάρα πολλές λεπτομέρειες και αυτό μας επέτρεψε να καταλάβουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος και τις απειλές. Η χώρα μου είναι η Πολωνία, η οποία δυστυχώς ε, έχει πληγεί από αυτή την αρρώστια, όπως φάνηκε και από το χάρτη. Εγώ είμαι από τα σύνορα. Ε, εκεί στις συνοριακές περιοχές έχουμε το πρόβλημα, αφορά μόνο κάποιες περιοχές συνοριακές, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές των χείριων προϊόντων της χώρας έχουν πέσει. Και βεβαίως οι χειροτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Έχετε πάρει πολύ αυστηρά μέτρα, πολύ μαξιμαλιστικά και έχετε στη διάθεσή σας ένα, μια πανοπλία μέσων που χρησιμοποιείτε πολύ καλά. Υπάρχουν και κίνητρα που δίνουμε στις ζώνες ε, που έχουν ε, πληγεί, όπου παροτρύνουμε τον κόσμο να μην ε, εκτρέφει χείρου για τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει με πλέον έξοδα. Πρόσφατα υπάρχει και ένας νόμος, ο οποίος έχει υιοθετηθεί για ε, την απειλούμενη περιοχή που δεν υπάρχει ακόμα η άρρωση, την Πολωνία εννοώ, δεν υπάρχει ακόμα η άρρωση, αλλά θα μπορούσε να προκύψει. Και που είναι γειτονική με την ε, πλήγησα περιοχή. Ε, Παραδείγματο χάρη, κάποιοι που είχαν αγοράσει χειρίδια, α πούμε, τα δώσανε σε ανθρωπιστικέ οργανώσει μετά. Όλα αυτά γιατί σα τα λέω, κύριε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά τα μέτρα, όλα αυτά τα επιπλέον ε, μέτρα που έχει ε, αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ θα τα χρηματοδοτήσουμε, θα τα πληρώσουμε το δικό μα προπολογισμό ή θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ε, συγχαίρω για την έκθεση. Αλλά όπως ε, είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, δεν, δεν αναφέρατε καθόλου την ε, Ιταλία. Ε, τη Σαρδινία συγκεκριμένα που υπάρχει μια εστία εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι Σάρδα. Εδώ και χρόνια Σαρδινία υπάρχει το πρόβλημα τη πανόλης των χείρων και πραγματικά με κατέπληξε το γεγονός ότι η Κομισιόν το ανέφερε στην παρουσίασή της. Παρά το γεγονός όμως ότι έχει γίνει έχουν γίνει παρεμβάσεις και από την ίδια Επιτροπή. Ήδη το 2013 είχε στείλει εκπροσώπους της Κομισιόν για να αξιολογήσει την εφαρμογή των μέτρων για την πανόλη των χείρων στη Σαρδινία. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί. Και λόγω της πρακτική πρακτικής που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα στην Ιταλία, όπου ζητάμε δηλαδή λεφτά από την Ευρώπη, χωρίς παρόλα αυτά να δώσουμε καμία συνέχεια. Χωρίς να εφαρμόσουμε δηλαδή τις κατάλληλες πολιτικές για τον περιορισμό της επιδημίας. Πρόβλημα λοιπόν με τα ταμεία, με τα λεφτά, αλλά όχι μόνο. Στην Ιταλία ποιος θα έπρεπε να ασχοληθεί, με την προστασία των ζώων. Ένας ε, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, μάλιστα έχει φτάσει, έχει φτάσει να τον ε, ελέγχει η δικαιοσύνη για μια ύποπτη υπόθεση με, με εμβόλια. Ε, ολόκληρη τομής λοιπόν ε, κτηνοτροφική βρίσκονται σε κρίση. Και ποιος την πληρώνει, οι τίμοι πολίτες. Είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να δοθεί μια απάντηση από την Ευρώπη. Επευκαιρία να σας πω ότι μέχρι τις 18 Οκτωβρίου υπάρχει μια task force η οποία επισκέπτεται την ε, Σαρδινία. Ο υπεύθυνο για την εποπτεία, για τη χρήση των ε, ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων υποτίθεται θα πρέπει να ελέγξει και τα προγράμματα. Ε, και το πώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται από τους ντόπιου, τους άρτους δηλαδή στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον κόσμο ότι η Task Force ελέγχει σωστά ε, το πώς ελέγχονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες διαβεβαιώσεις για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ κύριε Σουαζό. Και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η παρουσίαση αυτή, η παρουσίαση αυτή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ παθιασμένη. Και θα ήθελα να σχολιάσω όπως ο κ. Αγνιού ότι προφανώς το θέμα αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ανησυχεί τους εκτροφείς, ανησυχεί τους κυνηγού. Και θα ήθελα να μας πείτε με ποιο τρόπο, α, ποια τι συμπτώματα έχει η ασθένεια αυτή σε ό,τι αφορά τους αγριόχειρους και κατά πόσον θα μπορούσε να μεταδοθεί από άλλα ζώα, μέσω των αλεπούδων για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Και δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Ίσως θα μπορούσατε να πάρετε το λόγο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ετέθησαν για τους αγριόχειρους, γιατί είπατε ότι δεν θα υπήρχαν επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την σου αυτή, αλλά τι γίνεται με τους αγριόχειρους. Γιατί αυτό δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένο με το θέμα. για τις ε, διάφορες περιπτώσεις ε, βλέπουμε ότι δεν τηρούνται κάποια πρότυπα και κάποιες προδιαγραφές και αυτό προφανώς επηρεάζει με τη σειρά του και τους εκτροφείς. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους αγριόχειρους. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Πολλοί από εσάς ε, βλέπω ότι γνωρίζετε σε βάθος τα κτηνιατρικά ζητήματα. Χαίρομαι ιδιαίτερως. Να απαντήσω λοιπόν στις ερωτήσεις. Λίγο πολύ ε, με τη σειρά που ετέθησαν και θα καταλάβετε, ότι έχω και κάποια ζητήματα να τα απαντήσω όλα αυτά που με ρωτήσατε. Μία μεγάλη ομάδα ερωτήσεων έχει να κάνει με το τι κάνουμε με τους αγριόχειρους, τι κάνουμε με τη θηρευσή των θηλυκών. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά αυτά τα άγρια ζώα. Δύο εργαλεία έχουμε βασικά. Καταρχάς τα κίνητρα. Για να δοθεί κίνητρο τους ε, κυνηγούς να θηρεύουν θηλυκά, τους πληρώνουμε. Πληρώνουμε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα γενναιότερα πόσα. Δίνουμε μεγάλα πόσα για τους κυνηγούς, στους κυνηγούς για τα κουφάρια θηλυκών ζώων. Και στη συνέχεια το κουφάρι αυτό το καταστρέφουμε. Και αυτό συνδέεται με μεγάλο κόστο. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα κίνητρο για να προωθηθούν οι σωστέ ε, πρακτικές στο κυνηγή. Κάνουμε ενημερωτικέ εκστρατείε, λέμε στου ε, κυνηγού τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Και αυτό χρηματοδοτείται κατά 75% από το κοινωνικό προπολογισμό. Και σε τελική ανάλυση ενημερώνουμε και τις περιβαλλοντικές αρχές ποιες πρακτικές είναι αρνητικές. Όπως για παράδειγμα οι στοχοφατημένες, ε, το στοχοφατημένο κυνήγι που απαγορεύεται. Καθώς και η παραγή τροφής στα άγρια ζώα για να αυξηθεί ο πληθυσμός. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό στην παρούσα φάση. Άρα έτσι θεωρούμε ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά του αγριόχειρους είμαστε καλυμμένοι. Ξέρουμε πώς μεταδίδεται η ασθένεια. Δεν είναι καινούρια. Δεν ε, περνάει από τις μύγες, ούτε από τις αλεπούδες, ούτε από γήπες ε, και αρπακτικά πουλιά νεκροφάγα. Ξέρουμε τα μονοπάτια που περνάει η νόσος, γιατί έχουμε εμπειρία με την ασθένεια αυτή από το δεκαετία του 60, του 70, του 80 στην Ιβρυκή Χερσόνησο. Ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται και τι θα πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζονται εικασίε. Ξέρουμε τι έγινε στην Πολωνία το καλοκαίρι. Πολύ καλά. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της των δράσεων ενός ατόμου, ενός εγκληματία, ο οποίος διώχθηκε από την αστυνομία και ο οποίος πολλούσε τέτοια χειρίδια στην αγορά. Αυτό δεν ε, είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι ο εγκληματίας αυτός ε, έδρασε πολύ κοντά στη μολυσμένη περιοχή, αλλά αυτό θα μπορούσε να συμβεί και διασυνοριακά. Η ανθρώπινη συμπεριφορά προφανώς και το ανθρώπινο έγκλημα είναι καθοριστική σημασία και για να αντιμετωπίσουμε τις δραστηριότητε αυτέ, ε, φυσικά εδώ επισερχόμαστε σε άλλα λιμέρια πέρα από τα κτηνιατρικά ζητήματα. Τώρα πώς συνεργαζόμαστε με τους γειτονές μας. Με τους Ρώσους ομολογώ ότι σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή διαλόγου που... και των συζητήσεων ε, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και πλέον καλυπτόμεθα από το έργο και τους κανόνες των διεθνών οργανώσεων, όπως είναι η ΦΑΟ, η Παγκοσμία Οργάνωση για το Τρόφιμα. Έτσι λοιπόν δραστηριοποιούμαστε και Μιλάμε με τους Ρώσους και έχουμε αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα τα οποία σημειώθηκαν ε, κοντά στη Φιλανδία στη Ρωσία είναι ενσυχητικά αυτά τα κρούσματα. Τουλάχιστον μας ενημέρωσαν, είμαστε ενήμεροι και συζητάμε τα ζητήματα αυτά. Τώρα ποιε είναι τα προβλήματα στο ρωσικό σύστημα. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την ανάθεση κονδυλίων και την καταπολέμηση των ε, κρουσμάτων. Αλλά τουλάχιστον μα λένε πού βρισκόνται, που βρίσκονται. Με ειλικρίνεια. Η Λευκορωσία είναι άλλη υπόθεση. Αυτή είναι ακόμα στη φάση τη άρνηση. Λένε ότι δεν έχουν κανένα κρούσμα από το 2013 και μετά. Άρα, από πλευρά νομική και κτηνιατρική, θεωρούνται ελεύθεροι από οποιοδήποτε κρούσμα. Και εμεί υποτίθεται ότι είμαστε επικίνδυνοι. Και μα το λένε και κατάμουτρα. Μα λένε, Α, εμεί δεν έχουμε πρόβλημα. Εσεί φταίτε. Αυτό είναι γελίο. Είναι προσβολή. Κατάμουτρη πώς να συνεργαστεί κανείς με έναν εταίρο που είναι τόσο ανελικρινής. Δεν έβαλα στις διαφάνειες τον όρο εμβόλια, εμβολιασμοί. Είπα ότι κάνουμε έρευνα για να βρούμε νέα μέτρα για να ελέγξουμε την ασθένεια. Δεν τόλμησα να πω και να αναφέρω τα εμβόλια. Και γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ούτε καν υποψία εμβολίου στην παρούσα φάση. Από έχουμε παρασάγκας από το να έχουμε ένα υποψήφιο εμβόλιο το οποίο θα μπορούσε να περάσει από δοκιμές, το οποίο θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί και να περάσει ε, στην αγορά για τα επόμενα χρόνια. Μία, πολλά χρόνια. Δεν έχουμε, δεν έχουμε εμβόλια και πολύ απλά πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε την ασθένεια χωρίς εμβόλιο. Επενδύουμε βέβαια και στην ανάπτυξη εμβολίου. Αν υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα και προοπτική, θα το χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίω. Και θα προσαρμόσουμε την αντιμετώπιση μα. Σε κάποιε περιπτώσει ε, προτιμάμε και ένα περιορισμένη αποφωτικότητα ε, εμβόλιο, από, να μην υπάρχει καθόλου εμβόλιο. Αλλά δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, σα το λέω. Απασιόδοξα τα πράγματα. με ανησυχούν και οι χάρτες. Όταν κανείς παίρνει απόσταση και κοιτάει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την ασθένεια και αυτό είναι επιτυχές. Αλλά τώρα, σε ό,τι αφορά τα κουφάρια. Σε ό,τι αφορά την πανόλη των χείρων, έχουμε know-how, έχουμε τεχνογνωσία στην Ευρώπη. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι αντιμετωπίζουμε τα κουφάρια, τα επεξεργαζόμαστε με θερμική. αντιμετώπιση της μόλυνσης και ξέρουμε τι κάνουν οι χώρες που έχουν πληχθεί από την νόσο. Συγκεκριμένες τώρα ερωτήσεις από τη Φιλανδία. Πώς θα είμαστε πιο σίγουροι ότι τα στοιχεία που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε είναι έγκυρα. Πώς θα συλλέξουμε πιο αξιόπιστα δεδομένα και στοιχεία. Καταρχά να συνδεθούμε μαζί του, να συνομιλήσουμε μαζί του. Τα έχουμε προσπαθήσει όλα. Τι να σας πω. Και σε ό,τι αφορά του Ρώσου, πραγματικά σα το λέω με πάσα ειλικρίνεια ότι μα δίνουν σχεδόν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση του. Αν δεν έχουν αρκετά δεδομένα, ενδεχομένω αυτό να, φταί, να οφείλεται στο ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συλλάξουν πιο πολλά δεδομένα, αλλά το συναντάμε κάθε δύο-τρεις εβδομάδες. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης και είναι δύσκολο το θέμα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Το θέμα της διαπραγμάτευσης, ε, της ε, νομικής επίλυσης των ζητημάτων. Τώρα, κοιτάξτε, σε θέματα συνεργασίας τα πράγματα πάνε καλά. Τώρα, σε θέματα διαπραγματεύσεων δεν τολμώ να αποφανθώ. Και αυτό ξεπερνάει το δικό μου επίπεδο, αν θέλετε. Τα αγροκτήματα, πόσο θα πρέπει να μείνουν κενά προτού υπάρξει νέος πληθυσμός. Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε επακριβώς. Κάποιες εβδομάδες, μετά γίνεται μια δοκιμή, ένας έλεγχος για το πόσο καθαρό είναι το αγρόκτημα εισαγάγοντας ε, χειρίδια πειραματόζωα ουσιαστικά για να δούμε αν θα μολυνθούν. Μη σας ανησυχεί. Εδώ ξέρουμε επακριβώς τι πρέπει να γίνει και να σας πω ότι δεν είχαμε και προβλήματα στην Ιβρική Χερσόνησο. Το 1970 είχε μολυνθεί μισή Χερσόνησος και καταφέραμε τη δεκαετία του 80 να εξαλείψουμε την ασθένεια με πολύ πρωτόγονε μέτρα με θέματα ασφάλειας, υποχρεωτικά μέτρα ασφάλειας και απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ των εκτροφών, των αγροκτημάτων εκτροφής ε, χείρων και των αγριόχειρων. Άρα προωθούμε και δίνουμε κίνητρα για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και επιβάλλουμε και περιορισμούς. Αυτά τα δύο μέτρα ακολουθούμε. Και εδώ θεωρώ ότι η επικουρικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και κατά πάσα πιθανότητα οι χώρε οι οποίε έχουν μολυνθεί με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων ξέρουν τι μέτρα πρέπει να περάσουν για να περιορίσουν την ασθένεια για την βιοασφάλεια. Στη Μεγάλη Βρετανία είσαστε πολύ τυχεροί γιατί δεν έχετε σου γιατί Είχαμε και την κλασική πανόλη των χείρων πριν από 10 χρόνια στο Βέλγιο, στη Γερμανία και το καθεξής και κατάφεραν να εκριζώσουν την ασθένεια με εμβόλιο βέβαια. Αλλά η Αφρικανική Πανάλη των Χείρων είναι φιάλτη. Αν μία περιοχή όμω. δεν έχει αγριόχειρου, όπως η, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η Δανία, ειλικρινά δεν θα εισήγαγα αγριόχειρου σε αυτή τη φάση. Σαρδενία. σκόπιμα δεν ε, συμπεριλήφθηκε αυτό στους χάρτες που σας έδειξα. Γιατί δεν ήθελα να αναμίξω το πρόβλημα της Αφρικανικής Παναστοχήρων στην Πολωνία και στα κράτη της Βαλτικής με το πολύ γνωστό πρόβλημα της Σαρδενίας. Δεν ήθελα να προκαλέσω σύγχυση. Είναι διαφορετικά τα στοιχεία της ασθένειας. Και εδώ υπάρχει και φυσικά το κοινωνικό στοιχείο, πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό επίπεδο. Με πολύ προηγμένα κοινωνιολογικά ενδεχομένω μέτρα. Uh, και κάτι που δεν είναι μυστικό, υπάρχει και το στοιχείο της uh, τύχης, της εφαρμογής των βασικών κανόνων σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης. Τα ξέρουν όλα αυτά οι αρχές, ε, κάνουν ότι μπορούν, βελτιώνονται. Υπάρχει ένας αστυνομικός, ο περίφημος κομισάριο. Ε, υπάρχει και μια συγκεκριμένη αλυσίδα διοίκησης, η οποία εμπλέκει και την αστυνομία. φτιάχνει μια ολόκληρη πυραμίδα εξουσίας με σκοπό να επιληθεί ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι πρόβλημα λόγω της ανθρώπινης συμπεριφοράς ακριβώς. Προσπάθησα λοιπόν να μην μπλέξω τη Σαρδινία σε όλο αυτό, γιατί η Σαρδινία ευτυχώ, επειδή είναι νησί, α πούμε, περιοριστική αρρώστια και δεν αποτελεί απειλή η Σαρδινία για άλλου είναι πρόβλημα για τον εαυτό της. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά και εγώ και ο πρώην τμήματάρχης μου που είναι πάλι πίσω στη Σαρδινία και ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση της Σαρδινίας. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι το κοινωνικό στοιχείο στη Σαρδινία. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε και το μπαστούνι και το καρότο. Έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά από το Δαμείο Ανάπτυξη ε, Υπαίθρου, δηλαδή γεωργικά κονδύλια, για να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια αυτή. Είναι πολύ καλή αυτή η πρακτική και αυτό συνοδεύτηκε μάλιστα από ε, πίεση που ασκεί η αστυνομία. Πιέζεται και ο Δήμαρχο από την αστυνομία πούμε, για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμαρχο. Να εφαρμόσει τον νόμο, τον Ιταλικό νόμο και τον νόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά μεταξύ της κλασικής και της αφρικανικής πανόλης των χείρων είναι, απαιτεί πολύ προηγμένες ας πούμε κτηνιατρικές γνώσεις, γιατί οπτικά συμπεριφέρονται το ίδιο, αλλά η κλασική πανόλη ε, διαδίδεται πιο γρήγορα, μέσα σε μέρες σε μια κτηνιατρική εκμετάλλευση, ε, μέσα σε λίγες μέρες όλα τα ζώα είναι άρρωστα, ενώ η αφρικανική πανόλη έχει πιο αργή εξέλιξη. Γιατί, δεν απαντώ σε αυτό, η κλασική όμως πανόλη των χείρων πρέπει να πούμε ότι παρότι εξαπλώνεται πιο γρήγορα, σκοτώνει λιγότερο από την αφρικανική. Μετά από τρει-τέσσερι εβδομάδε, σε μία μολυσμένη εκμετάλλευση με αφρικανική πανόλη, τα περισσότερα ζώα είναι νεκρά. Ενώ για την κλασική πανόλη χρειάζονται μήνε για να αρρωστήσουν όλα τα. ή μάλλον αρρωσταίνουν γρήγορα, αλλά για να σκοτωθούν, για να πεθάνουν από αυτή την αρρώστια, χρειάζονται μήνε λοιπόν. Και παρότι μοιάζει το όνομα, πανόλη, πανόλη α πούμε, έχουμε, είναι διαφορετικέ αρρώστιε. Ε, για την κλασική πανόλη έχουμε ένα κλασικό εμβόλιο, αλλά δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Για την περίοδο επόση. γρήγορη είναι και τα, τα κλινικά συμπτώματα είναι πολύ εμφανή. Τα ζώα έχουν ψηλό πυρετό, απάθεια, δεν τρώνε και πεθαίνουν σε μέρες. Η πρόοδος από κτίριο σε κτίριο, πούμε, μέσα στην ίδια εκμετάλλευση, για να περάσει κανείς από τη μία, το ένα κτίριο πούμε, στο άλλο, η περίοδος επόσης συνολικά δεν είναι πάνω από μία εβδομάδα δηλαδή, για να εξαπλωθεί σε όλη, τη μεγα... σε όλη την εκμετάλλευση, εφόσον είναι μεγάλη εκμετάλλευση με πολλά κτίρια. Αλλά αυτό θα ξέρουμε, δεν είναι καινούρια η αρρώστια αυτή. Όλα αυτά είναι γνωστά, περιγράφονται και υπάρχει και η νομοθεσία η οποία είναι πολύ καλή για το πρόβλημα αυτό. Πολύ λεπτομερής, τα ξέρει όλα αυτά. Αχά, κάτι που ξέχασα. Οι επιπτώσεις στις τιμές, ε, βιωσιμότητα ε, και χρηματική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί να γλιτώσει χρήματα από τα κτηνιατρικά μέτρα ή από τα μέτρα στήριξη αγορά. έχουμε τελείως διαφορετικό πλαίσιο εδώ. Τα, τα κτηνιατρικά μέτρα, όλα αυτά που σας περιέγραψα δηλαδή σήμερα, χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς κανένα όριο για τα επιλέξιμα κόστη τα οποία είναι σημαντικά για τον έλεγχο της αρρώστιας. Πληρώνουμε, δηλαδή για τις ε, μολυσμένες ε, εγκαταστάσεις, πληρώνουμε για τις ε, εγκαταστάσεις που πρέπει να υποστούν πρόορη σφαγή και διακοπή της κτηνιατρικής δραστηριότητας. Πληρώνουμε για αυτό, πληρώνουμε όλες, για όλες τις δραστηριότητες για τους αγριόχειρους, για την καταστροφή των κουφαριών, για το, τη θύρα των θηλυκών αγριόχειρων, ε, όλα αυτά τα λέει η νομοθεσία και το ποσό συγχρηματοδότηση σε αυτήν την περίπτωση είναι 75%. Τώρα η ανάπτυξη άλλων και η χρησιμοποίηση άλλων ταμείων για να αντισταθμίσουμε τις τιμές της αγοράς ακολουθεί ε, τελείως λιγάκι διαφορετικό μονοπάτι νομικός πώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργοποιείται ανάλογα με τους παράγοντες της αγοράς από το κατόφλι που θέτουμε για τις τιμές της αγοράς. Δεν έχει να κάνει με την αρρώστια δηλαδή, είναι κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική, ένα διαφορετικό μέτρο. Δεν τα ξέρω εγώ, δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν ξέρω απ' έξω τις ε, αγορές τιμές. Νομίζω ότι απάντησα τις περισσότερες ε, ερωτήσεις, ίσως να ξέχασα κάποιες, αλλά δεν τα σημείωσα και όλα. Ούτε καν ε, και ο συναδελφός μου τα συμπτώματα στο, στους αγριόχειρους. Δεν τα βλέπουμε. Βρίσκουμε απλώς τα πτώματα, τα κουφάρια. Γίνονται θύματα, ας πούμε, αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, γιατί τα άρρωστα ζώα πριν πεθάνουν συμπεριφέρονται περίεργα. Περνάνε τους δρόμους, ή κάθονται και ξαπλώνουν πάνω στους δρόμους και τα σκοτώνουν τα αυτοκίνητα. Αν δέπετε μεγάλα ατυχήματα με, με αγριόχειρους, ε, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Μάλλον είναι άρρωστα, γιατί συνήθως δεν έχουν α, τάσεις αυτοχειρίας. Ελπίζω να σας άρκεσαν αυτά. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο να μιλήσει από την ε, πλευρά σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εκ μέρου των βουλευτών, πολλές ευχαριστίες. Με καθησυχάστε σε έναν βαθμό, γιατί είχα σκεφτεί ότι δεν ήμασταν ε, προετοιμασμένοι επαρκώ από άψη υποδομών για τέτοιε σοβαρέ επιζώτε. Πρέπει όμω σε κάθε περίπτωση να είμαστε προετοιμασμένοι, ο έννοιο. Η απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία φαίνεται τελικά υπεύθυνο αυτό που έκαναν, αλλά καταδικάστε από τι διεθνεί αρχέ. Μπορείτε να μου το αποσαφηνίσετε λίγο αυτό το θέμα. Well, at, at this point... Αυτή τη στιγμή το πήρα εκτός φαλούς. Βρισκόμαστε σε δίκη αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση της δίκης έχουν το δικαίωμα να κάνουν έφεση οι Ρώσοι στην έκθεση του πάνελ. Η έκθεση του πάνελ ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θέσης της. Αν το πάρουμε σαν ποδοσφαιρικό αγώνα θα έχουμε σκόρ 6 προς 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή έχει κερδίσει στα προκριματικά, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν είμαι δικηγόρος, μιλάω από την ιατρικής πλευρά Και είμαι αισιόδοξη γιατί βλέπω την ε, ποιότητα αυτό που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Στη Γενέβη, στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπου διεξάγεται η δική. Άρα είμαι αισιόδοξο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει την ημερήσια διάταξη, την έχουμε κλείσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινή συνεδρίσης, η επόμενη στι 7 και 8 Νοεμβρίου. Σας εύχομαι καλή επιστροφή. Σας ευχαριστώ και γεια σας